Ladies Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Καλώς ήλθατε στην ακρόαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διοικητικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλωσορίζω όλους τους παρόντες καθώς και τους συνομιλητές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε συνδεθεί, ελπίζω τουλάχιστον να είμαστε συνδεδεμένοι μέσω τηλεδιάσκεψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τον λόγο στην εισηγητή την κυρία Χαουτάλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ακόμη δεν έχουμε καθίσει όλοι. Αλλά ε, έχω τον χρόνο να καλωσορίσω και εγώ τον συνεισηγητή. Τον μόνιμο συνεισηγητή θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη σύγκριση για να εντοπίσουμε τις βασικές διαφορές και ενδεχομένω ομοιότητες μεταξύ των δύο επίρων. Ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση των τομέα αυτών είναι εξή. Η Ευρώπη Αμερική συνάπτουν όλο και στενότερους δεσμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, διαπραγματεύονται τη γνωστή TTIP για το εμπόριο και τι επενδύσει. Συμφωνία η Επιτροπή οποία ενδιαφέρεται τα μάλα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο με 12 επιτροπέ. Η συμφωνία δεν αφορά μόνο του δεσμού και τα τελωνία παλιά, αφορά την εναρμόνιση κανονιστικών μέτρων και διοικητικών διαδικασιών. Σήμερα λοιπόν δεν θα συζητήσουμε την TTIP και τις λεπτομέρειές της, όμως αυτά το οποίο θα συζητήσουμε αφορούν και τις συζητήσει για την TTIP. Μας ενδιαφέρει για παράδειγμα πως το διεθνές δίκαιο και άλλες διεθνείς συμφωνίες επηρεάζουν τις διοικητικές μας διαδικασίες. Κάτι άλλο που θέλω να σημειώσετε είναι ότι μπορούμε να μάθουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, παραδείγματι, όσον αφορά τον νόμο για την ελευθερία της πληροφόρησης. Πολύ πιο προχωρημένη νομοθεσία σε σχέση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή για την πρόσβαση στα έγγραφα. Η Επιτροπή μου ανέφερε σήμερα το πρωί να συγγράψω ένα κείμενο εργασίας όσον αφορά το θέμα σε συνεργασία με μαθα εργασίας, η οποία αποτελείται από μέλη και από άλλες βεβαίως πολιτικές ομάδες. Στις προηγούμενες εντολές εμείς πανεπιστημιακοί ιδρύματα και ούτω καθεξής. Έκανα πολλή δουλειά επί του θέματος. Θυμίζω τον κύριο Μπέρλιγκερ από την προηγούμενη μας θητεία και βεβαίω τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή για την καθιέρωση και βελτίωση των διοικητικών μας διαδικασιών. Ο στόχος απόψε είναι η συγγραφή μιας πρότασης τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το διοικητικό δίκαιο, στο οποίο θα ενσωματώνται οι καλύτερες καλές πρακτικές και προκειμένου όπως είπα έχουμε να μάθουμε πιστεύω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω ότι η σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί. Να ξεκινήσουμε. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ κυρία Χαουτάλα. Πριν ξεκινήσουμε να καλωσορίσω και πάλι τους προσκεκλημένους μας Θυμίζω ότι τα χρονικά όρια είναι στενά. Ξεκινούμε ούτως ή άλλως με καθυστέρηση. Θα είμαι αυστηρός με όλους ανεξαιρέτως. Παρακαλώ να τηρήσετε καταρχάς το όριο των 15 λεπτών για τη δική σας παρέμβαση. Ο καθηγητής Ματίας Goldman από το Εθνικό του Max Planck του συγκριτικού διεθνού δικαίου και διεθνού δικαίου έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, ελπίζω να με ακούτε. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου να σα απευθύνω το λόγο σήμερα. Σήμερα το θέμα μου δεν αφορά τη, την αμερικανική νομοθεσία, αλλά το τι μπορούμε να μάθουμε από το διεθνέ δίκαιο για τις ευρωπαϊκές διοικητικές διαδικασίες. Ελπίζω ότι η παρουσίασή μου θα σας βοηθήσει. Το θέμα είναι πώς επηρεάζει το διεθνές δίκαιο στην κωδικοποίηση των ευρωπαϊκών διοικητικών διαδικασιών. Ποιοι διεθνείς κανόνες λοιπόν ισχύουν και αφορούν τις διοικητικές μας διαδικασίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερεθνικό. Πριν από έναν αιώνα, το ερώτημα θα ήταν μάλλον αστείο, διότι το διεθνές δίκαιο αφορούσε μόνο τις διακρατικές σχέσεις κάτι το οποίο έχει αλλάξει εντελώς. Το διεθνές δίκαιο άπτεται πολλών ζητημάτων σήμερα, τα οποία απτώνται της ε, εθνικής αρμής Αυτό βεβαίω για τις επιπτώσεις του και στις διοικητικές διαδικασίες. Γενικώ υπάρχουν πολλοί κανόνες και νόμοι που αφορούν όπως είπα και άπτονται των εθνικών διοικητικών διαδικασιών. Δεν ξέρω τώρα πώς θα σας δώσω μια γενική επισκόπηση αυτών των κανόνων και των επιπτώσεών τους. Ένας, μια απλή επαρρύθμιση θα ήταν εξαιρετικά πληκτική. Σκέφτηκε λοιπόν να αναφερθώ στις γενικές αρχές. Αυτό κάνουν οι νομικοί όταν θέλουν να παρουσιάσουν κάτι με τρόπο συνεκτικό. Θεωρώ επίση ότι οι ευρωπαϊκέ διαδικασίε, διοικητικέ διαδικασίε μπορούν να ωφεληθούν από τι αρχέ, διότι οι αρχέ αυτέ μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικέ περιπτώσει. Για τον λόγο αυτών θα πω καταρχά λίγα λόγια για τη φύση και τη διαμόρφωση αυτών των αρχών και αμέσω εν συνεχεία θα παρουσιάσω πέντε διεθνεί βασικέ νομικέ αρχέ που πιστεύω ότι αφορούν τι ευρωπαϊκέ διοικητικέ διαδικασίε διευκρινίζω την έννοια αρχή. Δεν αποτελεί η πρόθεσή μου να πλήξετε με μια ομιλία περί νομικής θεωρίας. Γι' αυτό, θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο τύπους αρχών, δύο κατηγορίες αρχών. Γενικές αρχές του δικαίου, η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και αυτές είναι οι αρχές που βρίσκουμε σε διάφορες εθνικές ένωμες τάξεις. Είναι ένα λόγο που ξεκινούμε από τις εθνικές τάξει και το αμερικανικό δίκαιο όταν συζητούμε τις διοικητικέ διαδικασίε. Δεν είναι αυτό όμω το θέμα μας, γιατί θα έρθω μέσω στι άλλες αρχές που είναι οι αρχές του διεθνούς δικαίου. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Αναλύω καταρχά αν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία κανόν δικαίου που διέπουν τομείς ζητημάτων. Εάν διαπιστώσω ότι υπάρχει μια τέτοια κατηγορία, τότε μπορώ να συναγάγω ότι υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε αρχή. Φυσικά από τη μία περίπτωση στην άλλη οι αρχές αυτές δίνονται να διαφέρουν. Και εδώ ο καταλόγος με τις πέντε αρχές που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας μία προς μία. Οι αρχές αυτές βασίζονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές δικαιωτικές διαδικασίες του 2013. Εκεί αναφέρονται 10 αρχές, όμως ε, για λόγους συντομίας έχω συγκεράσει κάποιες από αυτές τις αρχές και έχω περιορίσει σε 5. Αναλογικότητα, νομιμότητα, έλλειψη διακρίσεων, δίκαιη διαδικασία, σεβασμός ιδιωτικότητας, διαφάνεια, ενημέρωση και το καθεξής. Για κάθε ε, μία από αυτές τις αρχές θα σας πω πώς αντικατοπτρίζονται, πώς άπτονται του σημερινού διεθνούς δικαίου. Αναλογικότητα αφορά τους λογικούς συλλογισμούς για την προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων. Είναι ένα βήμα το οποίο τα δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια κάνουν για τους σκοπούς της διαπίστωσης δικαιωμάτων. Πρόκειται για ουσιαστική αρχή, αλλά και διαδικαστική σημασία Πρόκειται για συλλογισμό και ο συλλογισμός βεβαίως είναι διαδικασία. Έτσι συνδέεται με τις διοικητικές διαδικασίες. Ποιοι είναι τώρα οι διεθνεί νομικοί κανόνε εν προκειμένου. Πολλοί από αυτού άπτονται τη αναλογικότητα. Είναι κριτήριο το οποίο πρέπει να ικανοποιούν, την αναλογικότητα δηλαδή. Ένα μεγάλο τομέα που μα ενδιαφέρει βεβαίω είναι το εμπορικό δίκαιο. Πολλοί κανόνε εμπίπτουν στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Το άρθρο 23 του οποίου, για παράδειγμα, τη παλιά ΓΚΑΤ προβλέπει εξαιρέσει από δασμού. Το ενδιαφέρον τη ΓΚΑΤ στο άρθρο 20 είναι ότι θεσπίζει δύο διαφορετικούς τύπους αναλογικότητας. Το ένα είναι η αναγκαιότητα και ο άλλος τύπος είναι ο απτόμενος, ο σχετιζόμενος με την αναγκαιότητα. Η πρώτη κατηγορία υπερτερεί σε ισχύ. Στην πράξη όμως η διαφορά είναι ελάχιστη και εν πολύς δυσδιάκριτη. Γιατί? Διότι το σχετικό το αρμόδιο εφετείο διευκρινίζει ότι ο τίτλος του άρθρου 20 της ΓΑΤ επιβάλλει στα κράτη ένα γενικό καθήκον καλής πίστης. Ενεργείας καλή την πίστη και αυτό αποτελεί ένα ενίο πρότυπο. Άλλες αποφάσεις από το χώρο του ΠΟΕ διαδικαστικοποιούν ούτως υπήν την υποχρέωση των κανόνων να πληρούν το κριτήριο της αναλογικότητας. Στην περίπτωση Homons, την υπόθεση Homons, κρίθηκε ότι οι εθνικοί κανόνες υπερτερούν των διεθνών στην περίπτωση, για παράδειγμα, αξιολόγησης κινδύνου. Και εδώ βλέπουμε την διαδικαστικοποίηση ουσιαστικά αυτού του κανόνα. Στο διεθνές δίκαιο η αναλογικότητα δεν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια. Τι είναι και που εφαρμόζεται. Η αρχή ε, πάντως θεωρείται γενικώ καθιερωμένη. Επίσης, η αναλογικότητα βρίσκει και πεδίο εφαρμογή στις συνθήκες για τα του ανθρώπου, όπου οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναλογικοί στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Εν τούτης, η νομολογία του δικαστηρίου, για άλλη μια φορά, έχει αποδυναμώσει τον κανόνα αυτόν από την ισχύ του διεθνούς προτύπου. Εν γέννη λοιπόν, η αναλογικότητα μπορούμε να πούμε παρόλα αυτά ότι είναι κατοχυρωμένη ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου. Όμως τα ωριά της δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα από τη μία νομιτάξη στην άλλη. Δύο είναι οι τάσεις. Η πρώτη είναι η τάση των δικαστηρίων να εναρμονίζουν την εξέταση αναλογικότητας ανεξαρτήτως του περιεχομένου. Η δεύτερη τάση είναι τα δικαστήρια να τείνουν να διατηρούν περιθώρια ευελιξία. Και μία τεχνική είναι η διαδικαστικοποίηση, όπως λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε την αναλογικότητα της αρχή, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ε, είναι αδύνατον βεβαίω να επιβάλλουμε απόλυτη πειθαρχία στα δικαστήρια, γιατί πάντοτε θα έχουν ανάγκη κάποιε ευελιξίε. Επόμενη αρχή, νομιμότητα, εξέλιξη διακρίσεων και θεμητέ προσδοκίε. Αυτά αφορούν ουσιαστικά την αντιμετώπιση τη αυθαιρεσία, την απαγόρευση τη αυθαιρεσία. Νομιμότητα λοιπόν σε διεθνέ επίπεδο. Πολλοί κανόνε λένε ότι οι περιορισμοί τη ελευθερία του ατόμου πρέπει να περιγράφονται και να προβλέπονται από νόμο. Κάποιε διατάξει περί δικαιωμάτων του ανθρώπου το τονίζουν αυτό, το ενισχύουν και ένα πρότυπο το οποίο έχει επεκταθεί με πολλού τρόπου. Πέραν όμως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ας πούμε το δίκαιο για τις διεθνείς επενδύσεις, ισότιμη δικαίη μεταχείριση και εκεί πρέπει τα μέτρα του χώρου, της χώρας υποδοχής να είναι αναλογικά. Όσον αφορά την καταρρίξη των διακρίσεων, την αρχή της μη διάκρισης, εδώ το δίκαιο είναι πιο κατακαιρματισμένο. Απαγορεύεται βεβαίως οι διακρίσεις, αλλά μόνο βάσει συγκεκριμένου δικαίου. Υπάρχουν διατάξεις για τις φιλετικές διακρίσεις, για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών κλπ. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες διατάξεις όμως. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά προχωρημένη, δεν έχει κάτι να μάθει. Όσον αφορά τις θεμητές προσδοκίες, η προστασία τους είναι μία από, τις βασικές, ένα από τα βασικά μελήματα της ρήτρα ισότιμης θεμητής μεταχείρισης. Σκοπός και εδώ είναι να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρότυπο. Δεν έχει γίνει όμως αυτό δυνατόν. Για να μην σας ε, ταλαιπωρώ, αυτό το οποίο αναμένουμε στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται το τρίτο είναι αλλαγή της πολιτικής του κράτους υποδοχής. Τώρα τι είδους αλλαγή πολιτικής. Κάποιοι λένε ότι είναι θέμα μάλλον αναλογικότητας, ότι δηλαδή τα κρατημέλη, κυβερνήσεις πρέπει να βρουν σε παραστάσεις, σε δηλώσεις που να ικανοποιούν τους επενδυτές. Και εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον πρότυπο, το οποίο όμως χρήζει περαιτέρω νομοθέτησης. Και αυτό θα συνιστούσε, αν προκειμένου. Ας περάσω τώρα στα θέματα δικαιοσύνης. Θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει γενικές εγγύησεις και <clears throat> συγκεκριμένες εξειδικευμένες εγγύησεις ως έχει εγγύα σε ένα γενικό επίπεδο <clears throat> δεν υπάρχει μια, ένας γενικός κανόνας της διαδικασίας. Αναγνωρίζεται όμως στη νομοθεσία και στις δικαιοδοσίες του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και αναφέρεται ότι η δίκαια δίκη η από πλευράς δικαιοσύνης πρέπει να θεωρείται ως γενική αρχή του διεθνούς δικαίου. Αν το εξειδικεύσουμε σε στενότερο πλαίσιο, μπορούμε να δούμε ότι για την υποστήριξη του δικαιώματος του να ακουστεί κανείς ε, ενώπιον δικαστηρίου αφορά όμως επίσης και θέματα εμπορικού δικαίου και έχει και διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή τη διτή χρήση. Το δικαίωμα να ε, εισακούγεται κανείς ε, σε σχέση με τα θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι κάτι εγγενές, ενώ διαφορετικά στο εμπορικό δίκαιο διαφοροποιούνται τα πράγματα βοηθά τα δικαστήρια και τους φορείς να ταυτοποιήσουν αν υπάρχει κάποιος ε, προστατευτικός σκοπός η ε, ανάγκη. Και με αυτές τις δύο διαφοροποιούμενες ε, διαδικασίες, αν δεν λαμβανόντουσαν υπόψη, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξειδικευτούν διαφορετικά, διότι για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου πολλές φορές ε, σε σχέση με άλλα θέματα μπορεί να υπάρξουν επικαλύψεις. Ε, τώρα, σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας, ε, της ιδιωτικής ζωής. Έχουμε και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά. Όμως ως προς αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο θεσπίζει διεθνείς προδιαγραφές και ας έρθω τώρα στην πέμπτη αρχή και τελευταία αρχή που θα ήθελα να αναφέρω, τη διαφάνεια, πληροφόρηση και διαβούλευση. Έχουμε δύο διαφορετικά στοιχεία αυτής της αρχής. Η πρώτη είναι ένα γενικό καθήκον, να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε σχέση με τα δημόσια έγγραφα για τους πολίτες. Το δεύτερο είναι πιο εξειδικευμένο καθήκον, συμμετοχής για εκείνους που αφορώνται άμεσα ή πιο εξειδικευμένα από κάποια ρύθμιση. Τώρα, για το πρώτο στοιχείο, τη γενική προσπελασιμότητα ως ε, δικαίωμα. Δεν υπάρχουν πολλά σε σχέση με αυτό στο διεθνές δίκαιο, εκτός από τον, την περιβαλλοντική νομοθεσία και την σύμβαση όρχους ε, της Δανίας. Και σε σχέση με το διεθνές δίκαιο υπάρχει σαφώς ε, η τάση, η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς διεθνών θεσμικών οργάνων, όμως ε, δεν έχει ακόμα αποκρισταλωθεί σε κάποια συγκεκριμένη μορφή ως αρχή. Και τώρα για το, την διαβούλευση υπάρχει ευρύ φάσμα όσον αφορά τα καθήκοντα ενημέρωσης και διαβούλευσης. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και καθήκοντα που εμπλέκονται όσον αφορά συμβάσεις ε, και συνθήκες ε, περιβαλλοντικές καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο ως προς αυτά ήταν αποφασιστική σημασία σε αυτά τα στοιχεία. Εδώ τουλάχιστον ε, ερχόμενοι σε σχέση με μια γενική αρχή, αν κάποιος αφοράται άμεσα από κάποια απόφαση με οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει καθήκον να γνωστοποιείται αυτό και να μπορούν να υποβληθούν και να διατυπωθούν σχόλια. Καταλήγω στο συμπέρασμά μου. Η διοικητική νομοθεσία έχει δύο ε, στόχους. Ε, αποτελεσματική διεκπαιρέωση των ε, διοικητικών καθηκόντων και διαφάνεια. Και πρέπει εδώ να δούμε την προστασία ατόμων κυρίως και όχι μόνο την αποτελεσματικότητα. Οι τελικές οι αρχές που αναφέρονται έχουν και μια ε, γενικευμένη διατύπωση. Αν πάμε σε συγκεκριμένες εξειδικευμένες λεπτομέρειες ε, δεν υπάρχουν ε, πολλά τέτοια συναφή στοιχεία εκτός από τα καθήκοντα που απορρέουν από συμβάσεις και συνθήκες. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι στην κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Προάγοντας αυτές τις αρχές μπορούν να προαθούν λοιπόν οι αρχές του διεθνούς δικαίου αντίστοιχα. Ευχαριστώ πολύ. We uh, Σας ευχαριστούμε εσάς καθηγητά. Τα επόμενα 15 λεπτά θα τα χρησιμοποιήσει η κυρία Ιωάννα Μέντες, Ιωάννα Μέντες από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη τη ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Οι επιπτώσεις ε, των διεθνών κανόνων στις ε, διαδικασίες στις διοικητικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το θέμα του ανοιχτού χαρακτήρα και της συμμετοχής και θα κάνω λόγο και κάποια προβλήματα απαριθμώντας κάποιες περιπτώσεις που θα φωτίζουν συγκεκριμένα το τι συμβαίνει και θα αναφερθώ στο τέλος και στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της ε, TTIP, της Διατλαντικής Σχέσης ε, Επενδύσεων και Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΕΕ. Το πρόβλημα γενικά. Τα θεμελιώδη ουσιώδη θέματα των διαφορετικών πτυχών της καθημερινής μας ζωής, της τροφής, ε, των τροφίμων που καταναλώνουμε, των φαρμάκων που καταναλώνουμε, των χημικών ουσιών κτλ. Όλο και περισσότερο αποφασίζονται από διεθνή ρυθμιστικά φόρα και μετά μέσω της ΕΕ. Οι διεθνείς υποχρεώσεις που εντάσσονται από πλευράς της ΕΕ μπορεί να έχουν διαφορετικές αρχές, μπορεί να είναι αποφάσεις διεθνών σωμάτων και φορέων σε σχέση με την κωδικοποίηση διεθνών συμβάσεων και συνθήκων που συμμετέχει και ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν τμήμα της νομικής τάξης πραγμάτων αλλά και αποφάσεις ε, φορέων και ε, σωμάτων που δεν έχουν ε, επίσημη διαφορετική άλλη βάση που εντάσσονται όμως σε διεθνείς θεσμούς στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας μέσω δηλαδή των οργάνων που αφορούν τη διοίκηση και βλέπουμε εδώ και το επίπεδο ακριβώς το διοικητικό που ε, εμπλέκεται είτε μέσω της ρυθμιστικής δράσης ε, των, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ ή των ίδιων των θεσμικών οργάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πύχης, ε, ως γνώμονας για να δούμε το πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί αυτή η δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η περίπτωση κατευθυντήριων γραμμών, προσανατολισμών κτλ. Όμως αυτοί οι κανόνες ε, το ότι εφαρμόζονται σε σχέση με την ΕΕ όπως και με τα διεθνή φόρα και οι τρόποι με τους οποίους ε, υιοθετούνται είναι ακριβώς ε, θέμα των διεθνών αυτών οργανισμών και υπηρεσιών. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Συχνά αυτό το ρυθμιστικό καθεστώς είτε έχει ρυθμιστική θεσμική βάση από πλευρά συνθήκων είτε όχι δεν έχει διαδικαστικούς κανόνες για την πρακτική εφαρμογή όλων αυτών όπως για άλλα θέματα υφίστανται στην ΕΕ και ταυτόχρονα οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΕΕ για την επεξεργασία αυτών των διεθνών κανόνων μπορεί να μην είναι εξίσου απαιτητική και αυστηρή όπως αν, είχαν, ε, αν χρησιμοποιούνται άλλες ε, βάσεις. Μέσω αυτών λοιπόν οι διοικητικές ε, διαδικασίες ακολουθούν ένα θα έλεγα ποικίλο πλαίσιο ε, ρυθμίσεων και αναφέρομαι στις διοικητικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις ε, που έχουν θεσπιστεί ως ε, πύχης και γνώμονας για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνώμονας και πύχης όσον αφορά την άσκηση των δημοσίων της δημόσιας δικαιοδοσίας και σε σχέση και με τα ίδια τα κράτη και μπορεί να ποικίλουν αυτοί οι κανόνες και ρυθμίσεις μπορεί να ε, έχουν ε, προσεγγιστεί για να επιλύονται προβλήματα αλλά και να δίνεται στους ενδιαφερόμενους πολίτες η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Εξαρτάται από το πώς έχουν σχεδιαστεί και προσεγγίζονται και αυτό είναι κέρια συνθήκη. Ανάλογα μπορεί κατά τη διάθεση τη ε, διαδικασία της ε, ε, λήψης απόφασης να διασφαλίζεται η ποικιλότητα, μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα της διασφάλισης της άσκησης εξουσιών. Δεν είναι όμως αυτός πάντα ο τρόπος με τον οποίο οι διαβουλεύσεις διεξάγονται. Όμως οι πρακτικές στην ίδια την ΕΕ και οι κανόνες ανοίγουν ένα δυναμικό, ένα πλαίσιο δυναμικού που μπορεί να εφαρμοστεί. Και αυτός ο ρόλος, ο συμμετοχικός για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε περιπτώσεις όπου η άσκηση των εξουσιών ε, αφορά και παραδοσιακά θέματα ελέγχου και βλέπουμε εδώ ότι σε σχέση με την αλυσίδα, ε, τον κρίκο της αλυσίδας αυτών των διαδικαστικών ε, διαδικασιών μπορεί να αφορά και εσωτερικούς ελέγχους ε, για να αυξηθεί η αυτονομία των εμπλεκόμενων και να δούμε κατά πόσον η νομιμότητα αυτών των πράξεων μπορεί να κατοχυρώνεται. Θα δώσω κάποια σύντομα παραδείγματα. Το πρώτο προέρχεται από την κοινή αλλιευτική πολιτική. Η ο ορισμός των ευκαιριών αλίευσης όπως και των ανώτατων επιτρεπόμενων αλιευμάτων είναι αποφάσεις που έχουν ευρύτατες ε, επιπτώσεις όσον αφορά τα, ε, τους όσους εμπλέκονται σε αυτή την πολιτική εσωτερικά υφίστανται τις, ε, στις διαδικασίες των συμβουλευτικών συμβουλίων όσον αφορά την αλλιευτική προσπάθεια, καθώς επίσης και από περιβαλλοντικές ομάδες και ομάδες καταναλωτών. Η διαβούλευση σε σχέση με όλα αυτά είναι κύριος πυρήνας σε σχέση με και τις δύο τελευταίες φάσεις της μεταρρύθμισης και πιο πρόσφατα το 2015. και η Ευρωβουλή επίσης έχει τονίσει τη σπουδαιότητα της διαβούλευσης με αυτούς τους φορείς και σώματα λαμβάνοντας υπόψη νομικές διαδικασίες πρέπει κάποια πράγματα να ληφθούν υπόψη όταν πρέπει να παρεκκλίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κάποιες ε, ε, αρχές πρέπει να δικαιολογείται αυτό να, υπάρχει, να υπάρχουν αντίστοιχα επιχειρήματα όμως επίσης και για την Επιτροπή Αλληλεία σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις που ε, συνεπάγεται η ευθύνη αυτή. Δεν ε, ε, ε, εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές αναλύωτα. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στην νομική τάξη πραγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρητά στο έγγραφο του 2006 εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ε, διαπραγματευτικές της ε, θέσεις ε, υπό το πρίσμα των διαδικασιών, των εγγράφων που αφορούν την κοινή αλλιευτική πολιτική για τις πολιτικές ευκαιριών αλλίευσης που πρέπει να προσφέρονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούνται αυτές οι αρχές από τα διεθνή σώματα και δεν είναι τόσο ανοιχτές όπως μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αυτό το οποίο θέλω να πω με όλα αυτά είναι ότι ενώ έχουν τις ίδιες επιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις αποφάσει, διότι εντάσσονται στη νομική τάξη πραγμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μπορεί να έχουν πιο ανοιχτό ή λιγότερο ανοιχτό χαρακτήρα, α, α, εξαρτώμενο αυτό το στοιχείο από το αν έχουν εσωτερικά υιοθετηθεί ή σε αντιστοιχεία με την διεθνή νομοθεσία. Το δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με τα φαρμακευτικά προϊόντα και αναφέρομαι κυρίως στις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων όσον αφορά την καταχώρηση φαρμάκων για χρήση στους ανθρώπους, το ICH. Το ICH είναι μια άτυπη διεθνής οργάνωση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών από τις Ηνωμένε Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Η EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατευθύνσει αυτέ γραμμέ είναι ουσιαστικά απαιτήσει τι οποίε πρέπει να ακολουθήσει η φαρμακευτική βιομηχανία κάθε φορά που προωθεί ένα νέο φάρμακο στην αγορά, κάθε φορά που κάνει αίτηση για μία νέα άδεια, προκειμένου να αποδειχθεί ότι όντω το φάρμακο είναι ασφαλέ. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε κατευθύνσει γραμμέ για τον τρόπο που δοκιμάζονται κάποια φάρμακα για την καταπολέμηση του καρκίνου, για παράδειγμα. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η ΕΜΕ, χρησιμοποιεί αυτέ τι κατευθύνσει γραμμέ για την αδειοδότηση συγκεκριμένων φαρμάκων. Θεωρείται ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν είναι λοιπόν δεσμευτικέ αυτέ οι κατευθύνσει γραμμέ, αλλά ακολουθούνται από την ΕΜΕ και ουσιαστικά καθορίζουν τη διαδικασία αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων. Στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα. Οι κατευθείαν γραμμέ ICH εγκρίνονται ακολουθώντα μια συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία συμμετέχει η EMA, αλλά δεν παρέχονται εγγύσει όσον αφορά την λεπτομερή ανάλυση όλων των παρατηρήσεων που υποβάλλονται, αντίθετα με αυτά τα οποία κάνει για παράδειγμα η EMA κάθε φορά που εξετάζει κατευθυντήρες γραμμέ. Η διαβούλευση ουσιαστικά λαμβάνει χώρα με διαφορετικό τρόπο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δεν εξετάζονται από την EMA, αλλά από τους εμπειρογνώμονες της ICH, χωρίς να δίνεται όμως περαιτέρω αιτιολόγηση ή περαιτέρω εξηγήσει για το τι ακριβώς διέπει τη διαβούλευση αυτή. Θεωρούμε λοιπόν ότι η EMA ως προς αυτό έχει περισσότερα χέγγια ασφάλειας ως προς την ανάλυση που κάνει. Επίσης, στα πλαίσια της ICH έχουμε επίσης και εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, Ενδεχομένως, λοιπόν να μην εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα συμφέροντα. Πάνω και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερα, η ενσωμάτωση των διεθνών αυτών αποφάσεων γίνεται με τους συγκεκριμένους αυτούς τρόπους και μπορούμε να δούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ενσωματώνται αποφάσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την νομιμότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όσα γίνονται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένω να μην ισχύουν διεθνώς. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις πιο ήπιοι κανόνες, λιγότερο ολοκληρωμένοι αν θέλετε κανόνες ή ακόμα και λυπή κανόνες μπορούν να συνάφουν περισσότερο με τις απαιτήσει που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ποια είναι η κάθε τη λεγόμενη επίπτωση των αποφάσεων αυτών. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες ε, αποφάσεις οι οποίες ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ισχύουν διεθνώς και ορισμένες, φορέ φορές οι κανόνες αυτοί οι οποίοι είναι άτυποι και δεν είναι δεσμευτικοί σε διεθνές επίπεδο αυτή τη στιγμή ενσωματώνται στο κοινοτικό δίκαιο γίνονται δεσμευτικοί. Και ουσιαστικά θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ρυθμιστικές αρχέ. Τελευταίο τώρα σημείο στην παρουσίασή μου να αναφερθώ στην συμφωνία TTIP. Εδώ τίθενται προκλήσεις διαφορετικού τύπου, διαφορετικά δηλαδή από όσα εξέθεσα μέχρι τώρα. Το κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με τη ρυθμιστική συνεργασία, με την υφιστάμενη μορφή που έχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν στα πλαίσια τόσο των νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη διακλαντική επίπτωση που μπορεί αυτοί οι κανόνες να έχουν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις αξιολογήσεις αντικτύπου, καθώς επίσης και στις ε, δεσμεύσεις διαβουλεύσεων, καθώς επίσης και στις ε, αξιολογήσεις αντικτύπου που ήδη έχουν ξεκινήσει. Πρόκειται λοιπόν για διαδικαστικές ε, υποχρεώσεις, οι οποίες δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή σε νομοθετικό επίπεδο. Την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δώσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις διαβουλεύσεις. Αλλά εφόσον εγκριθεί η συμφωνία TTIP θα μπορούσε όντως να προκύψει η υποχρέωση αυτή διαβούλευση και όντως θα μπορούσαν πλέον στα πλαίσια της TTIP να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες διαβούλευση. Και αυτό θα ήταν θετικό. Υπάρχει όμως μια σημαντική έλλειψη, ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι διαβουλεύσεις όπως προβλέπονται αυτή τη στιγμή στο κείμενο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την TTIP, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων αντικτύπου ή εν ώψη ενός μιας αξιολόγησης αντικτύπου. Και μάλιστα προβλέπεται συγκεκριμένο μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε πιο ποιοτικά ρυθμιστικά αποτελέσματα τα οποία θα είναι λιγότερα επαχθή για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και που θα προωθούν τη συνεργασία στα πλαίσια της TTIP. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, οι διαβουλεύσεις ενδεχομένως να μην αποτελέσουν φόρουμα φόρα μάλλον, στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν πολύ διαφορετικοί εμπλεκόμενοι και οι οποίοι θα μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους ή ακόμα και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως και ανεξάρτητα από την ανησυχία αυτή, θεωρώ ότι το σενάριο αυτό είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παρουσίασα πριν από λίγο. Αν όντω εγκριθούν έτσι τα πράγματα, τότε η TTIP θα εισάγει επισήμως συγκεκριμένου διαδικαστικού κανόνε διαβούλευση, οι οποίοι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή σε κοινοτικό ή διεθνέ επίπεδο. Το αν μας χαροποιεί αυτό ή όχι εξαρτάται, κανείς από, εξαρτάται από το πώς προσεγγίζει κανείς την διαβούλευση. Και ενώ το θεωρούμε ότι η διαβούλευση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μηχανισμό λήψης ποιοτικών αποφάσεων, όπως έχει πει άλλωστε πολλές σε πολλέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή, εφόσον ασπαζόμαστε την άποψη αυτή, τότε θα πρέπει να με αυτή την εξέλιξη. Πάντως, η διαβουλευση μπορει να αποτελεσει σημαντικο μηχανισμο ληψη ποιοτικων αποφασεων οπω εχει πει αλλωστε πολλε φορε η ευρωπαικη επιτροπη εφοσον ασπαζομαστε την αποψη αυτη τοτε θα πρεπει να ειμαστε χαρουμενοι με αυτη την εξελιξη παντω η συμμετοχη αυτη δεν θα πρέπει απλώ να περιορίζεται στα, σε μια απλή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει, να οδηγεί μια καλύτερη διακυβέρνηση. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει όντω να τρέφουμε και δικαιολογημένα θα τρέφουμε ανησυχίε. Είναι σημαντικό ότι εφόσον προχωρήσουμε σε αυτές τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις διαβούλευσης, τότε αυτές θα πρέπει αναγκαστικά να οδηγούν και συγκεκριμένες τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων τις συμφωνίες όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι συγκεκριμένοι κανόνες θα εγκριθούν και πώς θα επιβλέπονται αυτοί οι κανόνες. Ως προς αυτό λοιπόν η τύπη προβλέπει ένα μηχανισμό παρακολούθησης όσον αφορά την ρυθμιστική συνεργασία και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής όμως θα μπορεί και αυτός να αποφανθεί στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που εσωτερικά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. We Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να χαιρετήσουμε τους ομιλητές μας και να πούμε καλημέρα στην Νέα Υόρκη. Ο καθηγητής Richard Stewart από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης είναι μαζί μας και ετοιμάζεται να μας μιλήσει. Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα. Εδώ έχουμε ήλιο με δόντια όμως. Τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία η Επιτροπή σας υπέβαλε προς συζήτηση σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα από αυτά τα οποία μόλις προαναφέρθηκαν, από την Αμερικανική βεβαίως οπτική γωνία. Στο πλαίσιο πάντως της κανονιστικής μας εργασίας αφοτέλεθεν του Ατλαντικού. Σπέδω να δηλώσω ότι οι επιπτώσεις των διεθνών διαδικαστικών κανόνων στις αμερικανικές ε, διαδικασίες είναι ελάχιστες. Συνεπώς, κινούμεθα σε ένα σχετικά καθαρά εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι διεθνείς κανόνες δεν ε, απέτησαν δηλαδή τροποποίηση των δικών μας διαδικασιών. Είμαστε αρκετά ανεπτυγμένοι θα έλεγα σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά την ε, διαφάνεια, την συμμετοχή και την προσφυγή στην δικαιοσύνη. Με κάποιες εξαιρέσεις του διοικητικού οργάνου του ΠΟΕ στην υπόθεση Φρέμ Τέρτλ. Εκεί απαιτήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις κανόνων όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων και μεταποιημένων στο εξωτερικό προϊόντων. Τα πιο σημαντικά θέματα είναι αυτά τα οποία μόλις ανέφερε ο καθηγητής ο κ. Μέντες και αφορούν την εφαρμογή οδών διδικαστικών κανόνων που είναι αντικείμενο συμφωνία σε διεθνέ επίπεδο και φορούν όμω και από της τη εθνική ένωμη τάξη. Είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν οι εθνικέ διαδικασίε είναι σαφώ ανεπτυγμένε, όπω στι ΗΠΑ για παράδειγμα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι κανόνες είναι κανόνες που όπως είπα είναι σε εφαρμογή, συμφωνούνται σε διεθνέ επίπεδο, δεν έχουν ισχυρή τυπική ισχύ και εκεί προκύπτει το ζήτημα. Δηλαδή, το πώς ενσωματώνονται στην εθνική ενωμητάξη τέτοιοι κανόνες που δεν έχουν δοκιμαστεί παρκώς στην πράξη. Θα μιλήσω λίγο για τις επιπτώσεις που έχουν οι κανόνες μας, τις διεθνείς μας εργασίες, ιδιαίτερα εν ώψη της TTIP. Στο πλαίσιο δηλαδή της εργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διδικαστικών κανόνων. Αν εγκριθεί η TTIP όπως προτείνεται, διοικητικές διαδικασίες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα γίνονται όλο και οξύτερα όσο προχωρεί η συνεργασία μας. Όσο θα χρειάζονται δηλαδή διαπραγματεύσεις και θα τεθούν θέματα συμμετοχής και διαφάνειας προς το κοινό. Με δύο λόγια, να σας πω για τις σχετικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, το πώς προκρίνονται και θεσπίζονται αυτοί οι κανόνες στη χώρα μου. Οι σημερινές υφιστάμενε απαιτήσει για τους ομοσπονδιακούς οργανισμούς είναι κάθε φορά που θεσπίζουν ουσιαστικά νόμους να ενημερώνουν πρώτα απ' όλα, να εξηγούν τη βάση και τον σκοπό να αναφέρουν τις εναλλακτικές λύσεις και να είναι ανοιχτοί αυτοί οι οργανισμοί στις απόψεις ε, προσώπων ε, ΜΚΟ κλπ. Τα σχόλια αυτά μαζί με την τεκμηρίωση του προτείνοντος οργανισμού είναι δημόσια διαθέσιμα μεταξύ άλλων και στον ιστότοπο του οργανισμού και μετά από σχολιασμό εν τέλει ο οργανισμός θεσπίζει τον κανόνα συνοδευόμενο από την απαραίτητη υπεξήγηση. Σχολιάζει μάλιστα τις, ε, τα βασικά μελήματα και αντιρρήσεις. Σε αντιδιαστολή με την γενική αυτή πρακτική, και τόσο γίνεται στην Ευρώπη, οι δικοί μας κανόνες, εν γέννη, μπορούν να αναθεωρηθούν αμέσως και μετά την έγκρισή τους, την θέσπισή τους. για να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τα νομικά ζητήματα πριν ακριβώς αρχίσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες. Βάσει του νόμου για τις διοικητικές διαδικασίες οι κανόνες πρέπει να είναι λογικοί, αναλογικοί και τα δικαστήρια εξετάζουν πολύ στενά την αιτιολόγηση που δίνει ο οργανισμός για το συγκεκριμένο κανόνα κάθετος νόμος. Σταθμίζουν τα σχόλια του οργανισμού βάσει του υλικού που έχει συλλεγεί. Οι κανόνες αυτοί υπόκεινται σε δικηρική αναθεώρηση βασιντολών της εκτελεστικής εξουσίας υπό τους πρόεδρους Κλίντον και Ομπάμα είχαμε πολλές τέτοιε εντολές, αλλά και προηγούμενα επί Ρέγκαν και στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι αρχές της καλής νομοθεσίας βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών, να έχει προηγηθεί ανάλυση κινδύνου, ανάλυση κόστους, ωφέλειας και να υπάρχει δικαιολόγηση του σχετικού κόστους. Να έχει γίνει επαρκή ανταλλαγή απόψεων και να έχει υπάρξει επαρκή συμμετοχή. Και όλα αυτά βεβαίως στην περίπτωση που ο οικονομικός αντίκτυπος υπερβαίνει 100 εκατομμύρια δολάρια, τότε πρέπει να υποβληθεί και μια ξεχωριστή μελέτη επιπτώσεων. Όλα αυτά που βάλετε στο γραφείο του Κογκρέσου για τη διαχείριση του προπολογισμού πριν να δημοσιευθεί η τελική πρόταση για σχολιασμό. Μετά δημοσιεύεται ο κανόνα, η θετική ανάλυση, η έκθεση, η ανάλυση κινδύνου δημοσιεύεται και στον ιστότοπο του οργανισμού και αποτελεί μέρο ακριβώ του ψηφίσματο, του νέου νόμου. Το ίδιο δημοσιεύεται έκθεση του Γραφείου Διαχείρισης του Προπολογισμού. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στους ενδεχομένους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων. Το σύστημα αυτό αρχικώς επικρίθηκε από το Κογκρέσο και ομάδες καταναλωτών. Το σύστημα όμως αυτό έχει πλέον καθιερωθεί και πιστεύω ότι είναι ένα σοφό σύστημα, ένα ακρονίας λίθος της δικαιακής μας τάξης. Έχουμε δύο συστήματα διοικητικών αποφάσεων. Το ένα είναι το νομικό μας σύστημα βάσει του νόμου διοικητικών διαδικασιών που αναθεωρείται κάθε τόσο και το δεύτερο είναι το σύστημα ανάλυσης του διοικητικού μηχανισμού. Τα δύο αυτά επικαλύπτονται και τα δύο είναι επιδεικτικά, όπω είπα, αναθεώρηση. Γενικά θεωρώ ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι ούτε ο νόμο διοικητικών διαδικασιών, ούτε η διαδικασία διαταγών των διοικητικών αρχών διέπονται από πολύ συγκεκριμένου κανόνες. Οι κανόνε αυτοί δεν υπόκεινται σε διοικητική αναθεώρηση και εκεί οι συζητήσει μπορεί να είναι χρονοβόρες, όπως και χρονοβόρα μπορεί να είναι και η ανάλυση επιπτώσεων. Γι' αυτό και οι θέσει των διαφόρων μερών διατυπώνονται πολλές φορές με τρόπο και δεν είναι νομικά δεσμευτικέ. Και αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά ατόμων επιχειρήσεων, που θα θέλουν πολύ να γνωρίζουν ακριβώς τι ισχύει. Πρέπει να ξέρουν πώς ο τάδε οργανισμός εφαρμόζει τον τάδε κανόνα. Οι επικριτές επίσης ισχυρίζονται ότι αυτή η πληθώρα εγκυκλίων ούτως υπήν για να εφαρμοστούν τυπικοί κανόνες είναι προβληματική. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ασχοληθεί πολλές φορές με τέτοιου είδου περιπτώσεις. Και τώρα, πώς εφαρμόζονται διεθνείς κανόνες και πρότυπα στις ΗΠΑ. Προφανώς η διεθνής ε, συνεργασία παίρνει πολλές μορφές, έχουμε πολυμερείς διακυβερνητικούς οργανισμού που διατυπώνουν κανόνες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό των χωρών μας. Έχουμε διακυβερνητικά δίκτυα όπου εκπρόσωποι κρατών στο ICH, στην Επιτροπή της ε, Βασιλείας για τον τραπεζικό χώρο, όπως είπε και ο καθηγητής Μέντες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν μη τυπικές σχέσεις, ευέλικτες σχέσεις, υπάρχουν διμερείς επαφές, υπάρχουν συμφωνίε αμοιβέ αναγνώριση και ούτω καθεξής. Ένα πολυσχηδέ πλαίσιο. Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν στην εσωτερική ένωμη τάξη όταν συμφωνούνται τέτοιοι κανόνες στο πλαίσιο της διεθνού κανονιστικής συνεργασία. Ενσωματώνονται σε εθνικούς δεσμευτικού διοικητικού κανόνες. έχει τα πράγματα είναι σχετικά απλά, όλα αυτά υπόκεινται σε αναθεώρηση. Όμως έχουμε ένα ζήτημα για το οποίο έχω γράψει και το πει ο Πώς λειτουργούν αυτές οι διατάξεις, αυτές οι διαδικασίες πρακτικά όταν οι αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι για παράδειγμα έχουν συμφωνήσει ρυθμίσεις με τρόπο μη δεσμευτικό νομικά. Αυτό συμβαίνει διεθνώς και στην περίπτωση αυτή οι διαδικασίες δεν επηρεάζουν τόσο πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν οι λόγω κανόνες εφαρμόζονται μέσω γενικών κατευθυντηρίων οδηγιών, εγκυκλίων κλπ. Υπάρχουν εξαιρέσει βεβαίω όπου οι αμερικανικοί οργανισμοί έχουν αυξημένες εξουσίες βάσει της εθνικής νομοθεσίας να εφαρμόζουν κανονιστικές ρυθμίσεις που συμφωνούνται διεθνώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ας πούμε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Και εκεί υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής στην πράξη. Πολλές φορές αυτά γίνονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, άλλες φορές γίνονται μέσω μάλλον άτυπων διαδικασιών, εγκυκλίων και ούτω καθεξής. Και εκεί υπάρχει ευκαιρία συμμετοχή, αξιολόγηση από το κοινό, αναθεώρησης στα δικαστήρια, επανεξαίρεσης και αιτήσεις των οργανισμών για αιτιολογημένες απόψεις. Αυτά λίγο πολύ, αυτά είναι τα βασικά μελήματα, τα είπε και ο κύριος Μέντες. Για την TTIP τώρα συγκεκριμένα. Το πιο καινοτόμο στη της TTIP, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό το καινοτομό σύστημα κανονιστικής εργασίας, όπου εμπλέκονται πολλοί τομείς κανονιστικής δραστηριότητας. Θα δούμε αυτά κατά τομέα. Η TTIP προβλέπει διαρκή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθούν τα εμπόδια στο εμπόριο και για να προαχθεί καλύτερη νομοθεσία βάσει τεκμηρίωσης. ένας ε, ούτως πει μηχανισμός συντονισμού σε υψηλό επίπεδο θα είναι πολύ χρήσιμος. Ρόλο θα παίξουν επίση και οι γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή που υπόσχεται πολλά. Κύριε Καθηγητά, λέει ο συγγνώμη, ε, έχετε ήδη εξαντλήσετε 15 λεπτά, πότε θα σας παρακαλούσα να καταλήξετε στο συμπέρασμα. Πολύ ωραία. Με συγχωρείτε, φτάνω στο συμπέρασμα. Όπως προείπε ο πρόεδρος Ομπάμα. Εξέδωσε διαταγή για τη σχετική κανονιστική συνεργασία. Υπάρχει μια ομάδα εργασία εν προκειμένου έχουν γίνει και άλλες ε, καινοτομίε και γίνονται και άλλες και στην Ευρώπη. Αυτή λοιπόν θέλετε η πλατφόρμα, η θεσμική πλατφόρμα υψηλού επίπεδου συντονιστικού μηχανισμού από εδώ και πέρα φαίνεται ότι γίνεται μια πλατφόρμα για από κοινού αναλύση κινδύνου, από κοινού αξιολόγηση επιπτώσεων μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη συμμετοχή του κοινού με συντονισμό και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και για να κατακλείσω, στο αδερφό μου αναφέρομαι σε ένα σύστημα διαδικασιών, διαπραγματεύσεων, το οποίο έχει προτείνει ο παλιότερος Αμερικανός Ανώτερος Δικαστής, Boyd. Ένα πλαίσιο λοιπόν στο οποίο οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι εκπρόσωποι, η βιομηχανία, διαφορετικοί της οι καταναλωτές θα μπορούν πριν την θέσπιση κανόνων να προσυμφωνούν επί γενικών προσεγγίσεων και να χαράσουν και το δρόμο βάσει ανάλυσης κινδύνου και ανάλυσης κόστους ωφέλειας. Αυτό θα επιτρέψει λοιπόν στους κανόνες εκατέρθων του Ατλαντικού να προσεγγίσουν αμοιβαίως. Υπάρχει λοιπόν έδαφος για διαπραγματεύσεις, για αμοιβαία προσέγγιση και για λογοδοσία και συμμετοχή του κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Τα επόμενα 15 λεπτά είναι για τον κύριο Μαρέκ Γερεμπόφσκι από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Ε, not δεν έχουμε τις διαφάνειες, συγγνώμη. Okay, Θα ξεκινήσω λοιπόν, έστω. Χωρίς. Συγγνώμη, μπορούν οι τεχνικοί να διακόψουν τον ήχο που έχουμε από τη Νέα Υόρκη. Ας βλέπουμε την εικόνα, αλλά μην ακούμε τον ήχο, παρακαλώ. Chairman, members. Πρόεδρε, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να σας προσφωνήσω και να μιλήσω για τις διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ας ξεκινήσω με τη τη θέση ότι οι διαδικασίες οι διοικητικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τα κράτη-μέλη δεν έχει ενιοποιηθεί με κανέναν τρόπο. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας και δεν υπάρχει και κοινή προσέγγιση και αντίληψη για το τι εστί διοικητικές διαδικασίες. Κάποιοι θα έλεγαν ότι οι διοικητικές διαδικασίες αφορούν τις διαδικασίες π.χ. στην Γερμανία και αφορούν σε σχέση με ε, επιμέρους ε, υποθέσεις, οι ατομικές υποθέσεις. Άλλοι θα υιοθετούσαν την αμερικανική προσέγγιση ότι αφορούν δηλαδή τις ε, δραστηριότητες διοικητικών αρχών που όχι μόνο αφορά συγκεκριμένες δράσεις αλλά ε, καλύπτει και την νομοθεσία και τις ε, συμβάσεις ε, από πλευράς οργάνων της κεντρικής διοίκησης και τα λοιπά. Και όλα αυτά επειδή υπάρχουν, υπάρχει η διχοτόμηση σε σχέση με το ιδιωτικό δίκαιο και τις διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με τις ε, χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου, πράγμα το οποίο δεν ε, είναι το ίδιο σε σχέση με τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ένας κάποιος βαθμός ενιαίας αντιμετώπισης διοικητικών διαδικασιών. Αυτό στους τομείς, για παράδειγμα, που ρυθμίζονται ιδιαίτερα και σε μεγάλο βαθμό από την ε. Υπάρχουν και προσπάθειες κωδικοποίησης στοιχείων όσον αφορά την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, όσον αφορά το ψήφισμα του 2013, καθώς επίσης και τα όσα είπε η καθηγήτρια Μέντες. Και εδώ βρισκόμαστε πραγματικά στις, σε σχέση με το εκτελεστικό σκέλος σε σχέση με τις διατυπώσεις από πλευράς καθηγητών που αφορούν θέματα διοικητικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τώρα δημοσιεύονται και δημοσιοποιούνται στο ε, διαδίκτυο και θα δημοσιευθούν και σε άλλες γλώσσες ε, στο μέλλον. Ας επικεντρωθώ στην Πολωνία αυτή τη στιγμή. Μπορεί σε σχέση με την Πολωνία να ε, θεωρηθεί ότι υπάρχει ένας βαθμός κωδικοποίησης. Το 1928 υιοθετήσαμε τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες που είχαν αυστριακό πρότυπο. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που επηρεάστηκε από τις διοικητικές διαδικασίες της Αυστρίας. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην Τσεχοσλοβακία και πρώην Ιουγκοσλαβία κατά το παρελθόν και το ίδιο ίσχυε και για την Ουγγαρία. Ακόμα και μετά την ε, κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, παρόλα αυτά η νομική ε, επιρροή που είχε ασκηθεί εξακολουθούσε να υφίσταται. Και έχουμε λοιπόν και τον κώδικα διοικητικών διαδικασιών του 1960 που καλύπτει μόνο ατομικές πράξεις και αποφάσεις που ρυθμίζονται όπως ε, για παράδειγμα και ε, ε, από ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Η διοικητική αναθεώρηση, οι συμβάσεις οι διατάξεις, η χρήση διαφορετικών πληροφοριών καλύπτονται από διάφορες άλλες πράξεις. Ε, δεν διαφέρει λοιπόν πολύ η κατάσταση από το Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz της Αυστρίας, το γενικό δηλαδή νομικό νομοθετικό ε, διαδικαστικό πλαίσιο της Αυστρίας. Όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός κατακαιρματισμού και σε διαφορετικούς τομείς υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικοί κανόνες και κανονισμοί διαδικαστικοί. Υπάρχουν κεφάλαια όπως για παράδειγμα το κεφάλαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Χριστών Αρχών Διαχείρισης και Διακυβέρνησης. Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο ήδη ε, καλύφθηκε σε σχέση με το θέμα αυτό ε, συγκεκριμένοι κανόνες προέρχονται από έγγραφα για τα δικαιώματα του ανθρώπου ή αποφάσεις που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου ή για επιδιαιτητικές δράσεις όσον αφορά για παράδειγμα ε, επενδυτικές δραστηριότητες και αφορά ε, διοικητικές πτυχές διοικητικών θεμάτων. Υπάρχουν κάποια δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται αλλού όσο συγκεκριμένα στοιχεία διοικητικών διαδικασιών. Ξεκινάμε με το δικαίωμα του να εισακούγεται κανείς και να παρουσιάζει τα επιχειρήματά του. Ε, σύντομα, πολύ σύντομα θα υπάρξει μια αναφορά σε αυτά, αλλά πρέπει να πούμε ότι αν το δικαίωμα του να εισακούγεται κανείς αναγνωρίζεται παντού, ταυτόχρονα σημαίνει ότι η ίδια αρχή εφαρμόζεται ή πρέπει να εφαρμόζεται. Όμως στην ίδια την πραγματικότητα γίνεται διαφορετικά κατανοητό αυτό το δικαίωμα σε διαφορετικές χώρες ε, και περιοχές. Αλλού υπάρχει ένα στενότερο εύρος ερμηνείας, αλλού ευρύτερο φάσμα. Το δικαίωμα λοιπόν του να παρουσιάζει κανείς τα επιχειρήματά του και να, ε, ε, εισακούγεται που αναγνωρίζεται ως δικαίωμα στον, στη χάρτα των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα ευρύτερο τρόπο να γίνεται κατανοητό και να ερμηνεύεται. Κάποιος δηλαδή θα έχει δικαίωμα με αυτή την αρχή να προσφεύγει και να προστρέχει στις διοικητικές αρχές για ένα θέμα το οποίο εκρεμεί ή ε, τον ε, αφορά άμεσα. Τίθεται το ερώτημα ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει δικαίωμα να παρουσιάσει αυτά τα επιχειρήματα και να εισακούγεται. Μπορεί να αφορά αυτή η αρχή άτομο σε διαφορετικές περιπτώσεις ε, σε σχέση με, τους, ε, με τις διοικητικές αρχές ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε έναντι οποιασδήποτε διοικητικής αρχής. Υπάρχει λοιπόν μια ευρύτερη έννοια και ερμηνεία σε σχέση με αυτό το ε, δικαίωμα ως να αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε αφοράται από κάποια απόφαση έχει αυτό το, πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα και πολλών εμπλεκόμενων να παρεμβαίνουν. Θυμάμαι την περίπτωση κάποιου που ζούσε ένα χιλιόμετρο μα, μακριά από ένα τάξη και παρόλα αυτά θεωρείται ε, ότι και αυτός είχε δικαίωμα να εισακούγεται. Ε, υπάρχει λοιπόν ευρύτερο πλαίσιο ερμηνείας ε, για την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος. Τίθεται επίσης το ερώτημα τι βρίσκεται και πίσω από αυτό το δικαίωμα. Όχι ποιος έχει ένα τέτοιο δικαίωμα, αλλά τι πρέπει επίσης να συνυπάρχει ως συνεπαγόμενο. Διαρκής δηλαδή πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια και υποθέσεις από έναν ενδιαφερόμενο και η παρουσία του ίδιου αυτοπροσώπος όταν θα δι, ε, ε μαρτυρία ή τεκμηρίωση από κάποιαν αρχή. Επίσης οι αποφάσεις οι οποίες θα εκδίδονται από διοικητικές αρχές θα πρέπει να εκδίδονται μόνο όταν θα έχουν εισακουστεί οι εμπλεκόμενοι ενδιαφερόμενοι και θα έχει εισακουστεί η καταγραφή η άποψή τους ώστε να υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού και ε, ανταλλαγής επιχειρημάτων. Σε κάποιες χώρες αυτό λειτουργεί διαφορετικά δημοσιεύουν οι αρχές ε, ένα σχέδιο απόφασης ε, επί του οποίου σχεδίου μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους οι ενδιαφερόμενοι εμπλεκόμενοι. Υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, για αυτό το δικαίωμα όπως η αρχή της αμεροληψίας του αδέκαστου χαρακτήρα. Υπάρχει ένας σαφής κανόνας στην Πολωνία αν μια απόφαση έχει ληφθεί από μια αρχή ή από έναν άξιο ματούχο ε, χωρίς να υπάρχει αυτή η διασφάλιση αμεροληψίας ε, τότε θα πρέπει να απαλλάσσεται ή να αποπέμπεται ο υπάλληλος αυτός. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ευθύνε των αρχών έναντι αυτού του καθήκοντος είναι δεδομένες. Υπάρχουν και ε, περιορισμοί όσον αφορά διορίες και προθεσμίες. Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις της παραβίασης ή κάποιας παράβασης που μπορεί να διαπιστωθεί σε σχέση με τέτοιες ε, προθεσμίες ή διορίες, χρονικά όρια δηλαδή. Συγγνώμη, μια στιγμή σε σχέση με την παραβίαση ή παράβαση μιας τέτοιας χρονικής διορίας. Υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα τα οποία μπορούν να επιβληθούν σε σχέση με κάποιον αξιωματούχο. Πειθαρχικά δηλαδή να υποστεί τις συνέπειες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε εξουσιοδότηση. Δηλαδή θεωρείται ότι αν μετά από αίτημα δεν υπάρχει κάποια απόφαση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ε, κατά το οποίο πρέπει να εκδοθεί, ε, μπορεί τότε να ε, επιβληθεί κύρωση. Αυτό όμως δεν λειτουργεί πάντα διότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο η χρονική συνιστόσα η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά και η έγγραφη μορφή ή γραπτή μορφή ε, λήψης απόφασης ή δραστηριοποίησης από πλευράς ε, των αρχών. Έχουμε επίσης ένα σαφές ε, δικαίωμα το οποίο καθορίζεται για την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση των ενδιαφερομένων εμπλεκόμενων στο χαρτοφυλάκιο και τα στοιχεία εκείνα που τον αφορούν από πλευρά χαρτοφυλακίου. Δικαιώματα επίσης να γνωστοποιούνται τα στοιχεία για την απόφαση σε αυτόν τον εμπλεκόμενο. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να την χάνουν αυτή της πληροφόρησης, να έχουν αυτή την πληροφορία που θα τους διαβιβάζεται και να έχουν και τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή ε, για παράδειγμα έναντι της απόφασης αυτής ε, ακόμα και σε ακυρωτικό ε, δικαστήριο ή ανώτατο δικαστήριο. Και όλα αυτά απορρέουν ως τμήμα των διοικητικών αυτών διαδικασιών μέσα στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων. Καθώς επίσης και το θέμα των επανορθώσεων ή αποζημιώσεων που μπορεί να προβλέπονται. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα αποτελέσματα αυτού του πολύ ανεπτυγμένου πλαισίου διοικητικών διαδικασιών. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι δεν ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί, να μεταρρυθμιστεί ο κώδικας διοικητικών διαδικασιών. Και υπό την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να υπάρξουν κάποιες προσαρμογές όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική επικοινωνία, η ε, δυνατότητα να υπάρχει αυτή η επικοινωνία για όλους. Ε, ε, πράγμα το οποίο Έχουμε προσπαθήσει αρκετές φορές να το επιτύχουμε Έχουμε όμως και τομεακά εξειδικευμένη νομοθεσία όπου είναι πολύ έντονη η επιρροή της και αφορά επικεντρώνεται σε σχέση, με θέματα ε, μονοπωλίων όσον αφορά ε, κρατικές δικαιοδοσίες, ε, επιχειρηματικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες κτλ. Ας επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις υπάρχει ένα είδος σύγκρουση σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την εγγύηση των διοικητικών ε, αυτών ε, δικαιωμάτων. Γενικά απαιτείται χρόνος για να ε, λειτουργήσουν πλήρως όλα αυτά και κάποιου, κάπου θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Αναπτύσσοντας τέτοιες μπορούμε να ικανοποιήσουμε ε, τις αρχές που επιβάλλονται αμφωτέρωθεν. Όσον αφορά την Πολωνία τώρα, εμείς προχωρήσαμε και πήγαμε πολύ μακριά για να προστατέψουμε τα δικαιώματα των συμβαλωμένων εμπλεκομένων μερών σε σχέση με την, το παρελθόν. Το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ε, λήφθη υπόψη η διοικητική μεταρρύθμιση και σε σχέση με τις ε, φάσεις εφαρμογής ε, του διοικητικού δικαίου από τις αρχές, μέσα για παράδειγμα σε ένα χρονικό διάστημα πενταετές, πράγμα το οποίο καθιστά δυσχερές, για παράδειγμα, το να μπορέσουν με ταχύτερες διαδικασίες κάποια θέματα ε, ε, δημιουργίας αυτοκινητοδρόμων ή ε, οικοδομών ε, ή άλλων τέτοιων δομικών ε, εργασιών δεν μπορούν ιδιαίτερα να επιταχυνθούν. Πρέπει λοιπόν ένας ειδικό τομέας να ανοίξει και να θεσπιστεί ώστε σε σχέση με τα προνόμια κάποιων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες όπως τις τηλεπικοινωνίες και τις ε, ε, δραστηριότητες αυτές ε, να λαμβάνονται ξεχωριστά υπόψη. Έχουμε, θεωρήσαμε λοιπόν ότι υπήρχε σε ένα δευτερογενές επίπεδο αυτή η ανάγκη. Ανάγκη δηλαδή να εξεταστούν αυτές οι πτυχές ξεχωριστά και να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Παρότι έχουμε ένα καλώς ανεπτυγμένο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών, είμαστε υπέρ της κωδικοποίησης και ενιοποίησης ε, των θεμάτων αυτών όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο ένα θέμα δικαιωμάτων, αλλά είναι από την άλλη πλευρά και ένα θέμα του πώς θα μπορέσουν να ασκηθούν και να εγγυηθούμε την ε, ενάσκηση και εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων. Πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο Ιαν Χάρντεν, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Έχετε το λόγο κύριε Χάρντεν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας για τη διοργάνωση της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας ακρόασης. Σας ευχαριστώ επίσης για την πρόσκλησή σας, για τη δυνατότητα που δίνετε να μιλήσω για τις διοικητικέ διαδικασίες, καθώς επίσης και το άρθρο 298 και τη δυνατότητα μιας νομοθετικής πράξης διοικητικών διαδικασιών. Το άρθρο αυτό αποτελούσε καταρχάς μία νέα διάταξη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Στη συνέχεια, σχεδόν αυτολεξή, συμπεριλήφθη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού διαβάζουμε το ακόλουθο. Κατά την εκπόνηση της αποστολής τους, τα θεσμικά όργανα, φορείς, γραφεία και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την υποστήριξη μιας ανοιχτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο, οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να θεσπίσουν σχετικού ε, κανονισμού και σχετικέ διατάξει. Μέχρι στιγμή όμω κανένα τέτοιο κανονισμό δεν έχει θεσπιστεί που να έχει νομική βάση το άρθρο 298. Μπορεί ενδεχομένω όμως να δούμε τέτοιους κανονισμούς στο μέλλον. Γενικά έχει θεωρηθεί ότι το άρθρο αυτό πρέπει να έχει συγκεκριμένου περιορισμού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Θα ήθελα να κάνω δύο αρχικέ παρατηρήσει. Η ίδια διατύπωση, καθώ επίση και η ιστορία του άρθρου 298, καταδεικνύουν ότι αφορά μόνο την διοίκηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τη διοίκηση των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η διατύπωση αλλά και το γενικότερο πλαίσιο των συνθήκων προτείνουν ότι το άρθρο αυτό δεν αποτελεί νομική βάση για να ρυθμιστεί η σχέση μεταξύ θεσμικών οργάνων και προσωπικού τους. Μετά τις δύο αυτές αρχικές παρατηρήσεις θα ήθελα να επικεντρωθώ στο βασικό κατεμέ ερώτημα. Τι εννοούμε στο άρθρο 298 όταν αναφερόμαστε σε ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση. Θα αναφερθώ στις τρεις αυτές πτυχές ξεχωριστά αλλά θεωρώ και ελπίζω ότι θα γίνει σαφές ότι όλες αυτές οι πτυχές διασυνδέονται μία με την άλλη και υποστηρίζουν μία με την άλλη και από κοινού καταλήγουν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε καλή ή χρηστή διοίκηση. Μία ανοιχτή διοίκηση είναι αναγκαστικά διαφανής, δηλαδή το κοινό, καθώς επίσης και άτομα τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τη διοίκηση μπορούν να δίνει τι κάνει η διοίκηση, τι προτίθεται να κάνει, τι έχει ήδη κάνει. Μια ανοιχτή διοίκηση επίσης δίνει τις απαραίτητες ευκαιρίες για συμμετοχή στην διοικητική διαδικασία. Αυτά άλλωστε αποτελεί διαδικαστική δικαιοσύνη αν θέλετε ως προς τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην όλη διαδικασία αλλά και οι ίδιες οι συνθήκες αναφέρονται σε αυτό το δικαίωμα κάθε φορά που αναφέρονται στη συμμετοχή του κοινού, στη δημόσια συμμετοχή. Είτε αναφερόμαστε σε συμμετοχή ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στις αποφάσεις, είτε γενικότερα στη συμμετοχή του κοινού, πάντως σε κάθε περίπτωση τα ποιοτικά αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όσον αφορά την νομοθεσία. Ξέρετε ότι στο θεματολόγιο της πιο ευφυούς και αποτελεσματικής νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση Στόιμπερ αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις πλήρεις διαβουλεύσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η ποιότητα του νομοθετικού έργου. Ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα θεσμικά όργανα, ήδη προβλέπουν στα πλαίσια της πολιτικής τους και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων την δημόσια αυτή διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέπλεξε το κοινό σε μια γενικότερη διαβούλευση όσον αφορά την πολιτική που ακολουθεί για την διαφάνεια και μάλιστα άλλαξε το σχέδιο, το αρχικό σχέδιο κειμένου βάσει των παρατηρήσεων που είχε λάβει και στη συνέχεια είδε ότι ήταν τόσο σημαντικές οι παρατηρήσεις αυτές που έπρεπε να γίνει ένας δεύτερος γύρος διαβούλευσης και πάλι έγιναν επιπλέον αλλαγές προτού υποβληθεί ένα νέο κείμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά τη επίσης διαβουλεύεται ευρέω και πριν από δέκα περίπου χρόνια υπέβαλε ανακοίνωση όσον αφορά τις γενικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις κατευθύνες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθεί στη διαβούλευση με εμπλεκόμενα μέρη. Ο Ευρωπαίος Γεμεσολαβητής και το γραφείο του Ευρωπαίου Μεσολαβητή που είναι άμεσα υπεύθυνο για διαβουλεύσει αυτέ, περιλαμβάνει κάποιε προτάσει στην ιστοσελίδα του για το πώ θα μπορούσε η δημόσια διαβούλευση να συμβάλλει σε έναν μελλοντικό νόμο για τι διοικητικέ διαδικασίε. Τα όσα ισχύουν για τη συμμετοχή ισχύουν και γενικότερα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε νομοθεσίες που να διασφαλίζουν τόσο τα με μονομένα δικαιώματα των πολιτών στι διοικητικέ διαδικασίε και θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα υπέρ του δημόσιου συμφέροντο αυτών των διαδικασιών. Περνάω λοιπόν στη δεύτερη πτυχή τη χρηστή διακυβέρνηση, της ε, χρηστής διοίκησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 298, συγκεκριμένα στην αποτελεσματικότητα. Μία αποτελεσματική διοίκηση μειώνει τι απώλειε, χρησιμοποιεί του πόρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει όμω να θεωρούμε ότι όρος αποτελεσματικός στο άρθρο 298 περιορίζεται μόνο στα ζητήματα αυτά, ότι βέβαια είναι πολύ σημαντικά. Η διατήρηση, η τήρηση μάλλον αρχείων και μητρών μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική πτυχή της διοικητικής αποτελεσματικότητας και αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για ζητήματα διαφάνειας. Πιο ουσιαστικά όμως η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αναφέρεται και στον εξωτερικό αντίκτυπο που έχει η διοικητική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών κανόνων, καθώς επίσης και την διοικητική προετοιμασία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και με τη διαβούλευση έτσι και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει τους δικούς της διοικητικούς κανόνες προκειμένου να δει ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις που ενδεχομένω να έχουν στην πράξη κανόνες και πολιτικές που εγκρίνει. Αναφέρομαι προφανώς ε, στις γνωστές αξιολογήσεις αντικτύπου που ήδη ανέφερε η κυρία Μέντες. Ένας κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 298, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ένα πλαίσιο αρχών προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται καλύτερα οι εξολογήσει αντικτύπου στα πλαίσια της διοικητική δραστηριότητας. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα σε μία ακόμα πρόταση της ομάδας Stoiber. Η σύσταση παριθμών 9 στην τελική έκθεση προτείνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού σημείου επαφής όσον αφορά προτάσεις και όσον αφορά καταγγελίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Κατά την άποψή μου, ο στόχος της σύστασης αυτής θα μπορούσε να πληρωθεί καλύτερα μέσω μιας σύντομης διάταξης που θα μπορούσε να υπάρχει σε μια μελλοντική νομοθεσία διοικητικών διαδικασιών που θα υποχρέωνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά σε ετηρογημένα αιτήματα τα οποία μπορεί να στέλνει το κοινό και θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό άμεσης συμμετοχής, καθώς επίσης και ένα μέσο προώθησης της αποτελεσματικής διοίκησης. Το άρθρο 298 επίσης αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση ως ανεξάρτητη διοίκηση. Εκ πρώτη όψεω δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώ τι σημαίνει η έννοια αυτή. Σε άλλα σημεία η συνθήκη αναφέρεται σε ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητα θεσμικά όργανα, σαν ανεξάρτητους φορείς όπως οι κεντρικές ε, τράπεζες. Η διοίκηση όμως δεν αποτελεί από μόνη της ξεχωριστό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Άλλες διατάξεις ε, της ε, συνθήκης αναφέρονται σε συγκεκριμένους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου πάντως όρος ανεξάρτητος στο άρθρο 298 εκφράζει τις βασικές αυτές ιδέες που είχε εκφράσει ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής όταν αφέρθηκε στις βασικές αρχές των δημοσίων υπηρεσιών. Ότι ουσιαστικά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται προκειμένου να εξυπηρετούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τρόπο ώστε να προάγεται αυτός ο στόχος πάρουμε για παράδειγμα τις ομάδες επαϊόντων ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αληθεύει ότι τέτοιες ομάδες ε, ειδικών είναι όπως ε, και ε, λέσχες συζητήσεων ζητήματων. Επίσης αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει ποιου είδους εξωτερικές συμβουλές χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα καθήκοντά της να εκτελεστούν. Ωστόσο ο εξορθολογισμός δεν είναι το ίδιο <clears throat> όπως η τεχνοκρατία. Δεν υπάρχει τίποτα ανορθολογικό όσον αφορά την πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με την ε, εκτέλεση των ε, διοικητικών καθηκόντων. Υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα. Θεμητά όμω είναι ερωτήματα για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς ε, που διέπουν την λειτουργία τέτοιων ομάδων επαϊόντων. Πράγματι, ο Ομπουσμαν κάνει και μια εξέταση ξεχωριστή από πλευράς του για αυτό το θέμα και όλες οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διατάξεις, όχι μόνο όσον αφορά ομάδες επαϊόνων αλλά και ηθικά θέματα όπως ε, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα καθώς επίσης ε, και τις αρχές και την αντιμετώπιση θεμάτων λομπίστων και ομάδων πίεσης. Πρωτού ολοκληρώσω σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε, μια θεμε, σε ένα θεμελιώδες ερώτημα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία επιδικητικών διαδικασιών, ναι ή όχι. Ένα σημαντικό μέρος των νομοθετικών διαδικασιών σε σχέση με αυτές τις ε, διοικητικές διαδικασίες ήδη υφίσταται σε σχέση με τομεακά συγκεκριμένες ρυθμίσεις καθώς επίσης και γενικές αρχές ε, όσον αφορά την νομολογία του δικαστηρίου ή τις αρχές που ταυτοποίησε και εντόπισε ο καθηγητής Γκόλμαν σε σχέση με τις ε, περιπτώσεις και την ομολογία του ε, ε, δικαστηρίου. Άλλες, άλλα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά και την συμμετοχή στην σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ήδη εποφελούνται από εθελοντικές διατάξεις που υπάρχουν και μπορούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν και κάποιες δεσμευτικές αποφάσεις σε σχέση με αυτές τις πτυχές. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει και να πει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Επίσης θα μπορούσε να επιχειρηματολογηθεί ότι τέτοιου είδους ανεπάρκειες ε, με κατακαιρματισμένο ή εμβαλωματικό τρόπο πολλές φορές αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα θέματα τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, η συνθήκη είναι εκείνη η οποία ζητεί και πρέπει να απαιτείται έναν ανοιχτό τρόπο διοικητικών διαδικασιών και χρησιμοποιεί και συγκεκριμένη ορολογία διατυπώνοντας αυτά τα αιτήματα. Δεύτερον, νομοθετώντας υπό το πρίσμα του άρθρου 298 θα δώσει στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο, καθώς επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις γενικότερες αυτές ε, συνθήκες όσον αφορά τις ε, διοικητικές διαδικασίες και διατάξεις. Τρίτη και τελική, τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να αναφέρω απορρέει από τη δεύτερη παρατήρηση. Οι διοικήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διοικητικά της στοιχεία πολλές φορές ε, ε, χαρακτηρίζονται άδικα βέβαια σαν ένα είδους ε, τέρας που έχει την έδρα του, το λιμέρι του στις Βρυξέλλες. Όμως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδείξουν τη δική τους βούληση να συμμετάσχουν σε ένα ανοιχτό χαρακτήρα πλαίσιο διοικητική διαδικασίας και εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμητοποιώντας έτσι και νομιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των πολιτών της. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Γενικέ Γραμματεύ. Και τώρα ήρθε η χρονική στιγμή για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ερωτήσεις από τους Ευρωβουλευτές προς τους ε, εξέχοντες ε, ομιλητές που συμμετείχαν. Ελπίζω ότι είμαστε ακόμα σε επαφή με τον καθηγητή κύριο Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορεί και εκείνος να, παρακολουθήσει και να ακούσει τις διατυπώσεις των ερωτήσεων που ενδεχόμενα ίσως απευθύνονται και στον ίδιο εκείνον. Όμως φοβούμαι ότι μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να γίνει. Θα πάρουμε τις ερωτήσεις και μετά εσείς θα έρθει η σειρά σας ευμενώς να απαντήσετε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω σε σχέση με την TTIP, τη Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων με τις ΗΠΑ και τις ε, ΕΕ, σε σχέση με τη ρυθμιστική συνεργασία. Αν κατάλαβα καλά όλη την όλη συζήτηση για την TTIP, πρόκειται για αυτά τα θέματα κυρίως επίσης και για το ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σώμα ρυθμιστικής συνεργασίας μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης όπου αμοιβαία, αμφίδρομα θα μπορεί να εξεταστεί. Υπάρχει μεγάλος μικροφωνισμός και δεν μπορούν οι διερμηνείς να παρακολουθήσουν. Υπάρχει έντονος μικροφωνισμός και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον ομιλητή. Κύριε Κώστα, την ερώτησή σας προς τον καθηγητή Στιούαρτ τη στρέφεται ή όχι. But, uh, Ναι, και στον καθηγητή, αλλά νομίζω καλύτερο θα ήταν να στραφεί η ερώτηση να απευθύνεται και προς όλους τους συμμετέχοντες. Το λέω γιατί υπάρχει αυτός ο μικροφωνισμός. Yeah. Uh, Υπάρχει πρόβλημα σε σχέση και με τους διαρμηνείς επίσης με αυτό το μικροφωνισμό. Uh, let us wait for a Ας περιμένουμε ένα λεπτό ίσως για να αποκατασταθεί η επαφή ίσως αν γίνεται. Professor Stewart, do you hear us? Σας ακούτε καθηγητά Stewart. Σας ακούω τώρα, πιο πριν όχι. put up, uh, Τώρα σας ακούω. So I'm, I'm with you now. Δεν έχω εικόνα, αλλά όμως σας ακούω. We are taking the first... Τέλεια. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν διατυπώνεται και θα ακολουθήσουν όλες οι ερωτήσεις που θα πρέπει να ε, θέλουν να διατυπώσουν οι ευρωβουλευτές και όλοι οι όσοι συμμετέχουν ως ε, πραγματογνώμονες θα κληθούν να απαντήσουν. Κύριε Κώστα, την ερώτησή σας παρακαλώ. Η ερώτησή μου λοιπόν. Η ερώτησή μου αφορά την TTIP, Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τη ΣΥΠΑ και την ΕΕ και το σώμα ή φορέα ρυθμιστικής συνεργασίας. Υπάρχει ο στόχος και η πρόθεση νομοθετικά, νομοθετικές προτάσεις στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ να εντάσσονται σε αυτό το φορέα και να εξετάζονται από αυτό το φορέα νομοθετικά και ρυθμιστικά αν ενδεχόμενα θα δημιουργούσαν πιθανά εμπόδια ή προσκόμματα εμπορικά στις σχέσεις μεταξύ ΙΠΑ και ΕΕ. Κατά πόσον αυτό μπορεί και είναι συμβατό και συνάδει με νομικές αρχές ή όχι. Μήπως υφίσταται ο κίνδυνος εδώ η δημοκρατία να γίνει προσάρτημα των αγορών και να κινηθούμε προς μια δημοκρατία η οποία θα συνάδει με τις αγορές και μόνο και δεν θα είναι αυθύπαρτη αυτοτελής δημοκρατία που θα βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά το ελεύθερο εμπόριο θα έχει το πάνω Αυτό θα έλεγα εγώ είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό ως προοπτική. Μας ανησυχεί ως ενδυνάμει εξέλιξη και σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη πραγμάτων που θα μπορούσε να υφίσταται σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την ΕΕ. Ευχαριστώ. Any other questions? Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Mrs. Hautala. Η κυρία Χαουταλά. Um, Έχουμε μερικά λεπτά για γενικότερε παρατηρήσει, αλλά μεταξύ να ρωτήσω των Για τον μηχανισμό που περιέγραψε ο κύριος Στιούαρτ που θα είναι ενδεχομένω ο βέλτιστος τρόπος συντονισμού των κανονιστικών ζητημάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον εφαρμοστεί η TTIP. Θέλω να καταλάβω αν πραγματικά μιλάει για έναν υψηλό επίπεδο πολιτικό μηχανισμό, ο οποίο βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί και σε χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο. Το βασικό που ακούσαμε ήταν ότι πρέπει να υπάρχει προγενέστερη διαπραγμάτευση. Κύριε Μέντε, προβλέπετε, βλέπετε ότι ένα τέτοιο μηχανισμό μπορεί να ιδρυθεί, να δημιουργηθεί και ότι θα έχει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Άλλε ερωτήσει, παρακαλώ. Όχι. Κύριε Μέντε, μήπω ε, θέλετε να δώσετε μια πρώτη απάντηση. Ναι. Δεν γνωρίζω τι λεπτομέρειε τη ε, πρόταση του καθηγητού Στιούαρτ, αλλά από όσα άκουσα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σημερινή ευρωπαϊκή πρόταση. Για να υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο μηχανισμό κανονιστική εργασία. Υπάρχουν όμω βάσιμε ανησυχίε όσον αφορά αυτού του ρυθμιστικού φορεί. Ξέρω ότι γίνονται συγκεκριμένε προτάσει ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ επίση και του ε, Αμερικανικού Γραφείου ΟΙΡΑ. Το σώμα αυτό, ο φορέας αυτός θα επιβλέπει τις διοικητικές ε, διατάξεις που θα πρέπει να διέπουν τη συμφωνία TTIP. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η σύνθεση του φορέα αυτού και να δούμε αν τελικά ο φορέας αυτός θα πρέπει να απαρτίζεται μόνο από υψηλόβαθμους πολιτικούς αξιωματούχους ή αν θα πρέπει ο φορέας αυτός να είναι λίγο πιο ανορθόδοξος και να εμπεριέχει τελικά και ομάδες διασύνδεσης με βουλευτές. Αυτό ενδεχομένω να θεωρηθεί κάπως ανορθόδοξο, αλλά θα μπορούσε και αυτό να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της όλης συζήτηση που γίνονται για το μηχανισμό αυτό που θα μπορούσε να συμπεριλάβει ο TTIP. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη ε, εξέλιξη στον TTIP αν λάβουμε υπόψη μας τα όσα πρότεινε ο κύριος Στιούαρτ, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τη νέα αυτή θεσμική πλατφόρμα που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και τι διασύνδεση θα υπάρχει ανάμεσα σε αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την πλατφόρμα αυτή και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται παραδοσιακά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα όργανα της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε. Ενδεχομένως θα πρέπει τώρα να θέσουμε και το ερώτημα αυτό στον κύριο Στιούαρτ. Μήπως να πάρει το λόγο ο κύριο Στιούαρτ. Σας ευχαριστώ. Μ' ακούτε καταρχάς. όσον αφορά την εμπειρία που έχουμε στι Πολιτείε για τι διαπραγματεύσει αυτές τις ρυθμιστικές. Θα μπορούσα να σας στείλω ένα συγκεκριμένο άρθρο που έχει γράψει ένας ειδικό βάσει της εμπειρίας που έχει όταν ήταν ε, επικεφαλής του ναι. Συμβουλίου που είχε δημιουργήσει ο George W. Bush. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, ναι. πάλι υπάρχει ένα θέμα με τη διερμηνία. Δεν ακούμε καθόλου τη δερμηνία προς τα γαλλικά, λέει ο Πρόεδρος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Uh, so, uh, Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο θόρυβος. Λαμβάνουμε πολύ θόρυβο. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο αργά και καθαρά. Έλεγα ότι μια παρόμοια εμπειρία είναι η νομοθεσία και οι κανονισμοί για τη βενζίνη, την αναδομημένη βενζίνη, κάτι το οποίο έχει ενεργειακές αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βιομηχανίες, ε, κατανοητές, ε, μικιό, πυρογνώμονες, πριν θεσπιστούν οι κανόνες, κάθισαν γύρω του τραπέζι και το πράγμα εξελίχθηκε εξαιρετικά ομαλά προς ικανοποίηση των όλων. Το θέμα είναι πώς εξάγει αυτήν την διαδικασία ή μια παρόμοια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, στην διατλαντική σχέση, όπου έχουμε δύο διαφορετικές ένωμες τάξεις, η μια παρομοια διαδικασια εν παση περιπτωσει στην διατλαντικη σχεση οπου εχουμε δυο διαφορετικες ενωμες ταξεις η μία με τους δικούς της μηχανισμούς λήψη αποφάσεων. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική καινοτομία, αλλά όπως είπε η κυρία Μέντε. θα μπορούσε να είναι κάτι σαν αυτό κάποια εν μάλλον άτυπη διαδικασία που θα μπορούσε να εμπνέεται από τις κείμενες διαδικασίες στις ε, εθνικές ένωμες τάξεις. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο καθώς θα προχωράει και η TTIP επί αυτού του σημαντικού θέματος. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ. Και οι τρεις ε, αναπομείνοντες ε, καλεσμένοι θέλουν να σχολιάσουν. Ο καθηγητής Γκόλμαν πρώτα απ' όλα. Να μιλήσω γερμανικά μπορώ. Εντάξει. Και την ερώτηση του κυρίου Κέστερ να την απαντήσω αν γίνεται. Καταρχήν, συμμερίζομαι απόλυτα τις επιφυλάξεις σας. Υπάρχει πράγματι κίνδυνος δημοκρατικά ένας μη υπεύθυνο φορέας σε πολιτική εξουσία να ασκήσει υπερβολική ε, επιρροή ή εξουσία από πλευρά του. Ωστόσο υπάρχουν και καλά μαντάτα ή τουλάχιστον κάποια παρηγοριά. Παρηγοριά μόνο ένα. Υπάρχουν ήδη τέτοιοι φορείς και σώματα σήμερα ήδη και γι' αυτό υπάρχουν και προδιαγραφές για την λειτουργία τους. Και ο καθηγητής Στιουαρτ, η συνάδελφος ε, κυρία καθηγήτρια Μέντες και το Max Planck Ίδρυμα στην Χαϊδελβέργη εργάζονται εκ του σύνεγγης στην ε, εκπόνηση προδιαγραφών για τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την λογοδοσία, accountability και να γίνει κάτι καλύτερο και αποτελεσματικό. Τι κανείς και ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος ή καλός όσο ένα κοινοβούλιο. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε κάποια πράγματα να τα βελτιώσουμε. Δεύτερη, ε, δεύτερη καλή είδηση η εναλλακτική δυνατότητα για τεχνικές, τεχνοκρατικές τέτοιες δυνατότητες υπό ιδιωτικό πλαίσιο ρύθμισης ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πλαίσιο και ε, ιδιωτική, ιδιωτική πτυχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ προσεκτικά πρέπει να σταθμίσει το Κοινοβούλιο και σε λεπτομέρειες αυτά τα προβλήματα μπορεί να απαμβληθούν. Έστω σε κάποιο βαθμό μπορεί να μειωθούν. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ ο καθηγητής Διασμεμπόφσκι. Συμφωνώ. Η γενική αντίληψη περί κανονισμού στις πολιτείες είναι πολύ γενική. να σας πω είμαι ειδικό σε θέματα χρεογράφων. Η σχετική νομοθεσία, να ξέρετε, στον τομέα έχει εκπονηθεί από αμερικανικούς οργανισμούς. Και αυτό θα διαπιστώσουμε φοβούμε ότι είναι πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τώρα επειδή γνωρίζω την πολιτική πραγματικότητα στις Ηνωμένε Πολιτείες, ξέρω ότι υπάρχουν πολύ στενοί δέσμοι μεταξύ οργανισμών και του Κογκρέσου και ούτω καθεξής. Αυτοί οι δεσμοί εν της συνθήκης ε, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά ισχυροί. Συμφωνώ λοιπόν. Γενικό ε, Γραμματέα, ο κ. Χάρντεν. Πρόεδρε, η εμπλοκή του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή στην ε, περιορίζεται σε θέματα διαφάνειας, διαφάνειας των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε επισέλθει στην ουσία των θεμάτων. Η, προ... επάνηση λοιπόν, μου, λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι ε, προσωπική, αν θέλετε, και δεν είναι επίσημη θέση των οργάνων. Σύμφωνα με τον καθηγητή Goldman, ότι υπάρχει εμπειρία με κάποιο του διεθνέ κανονιστικό δίκαιο και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά ξαφνικά μόνο την TTIP. Δεν προκύπτει για πρώτη φορά δηλαδή η ανάγκη να συγκεράσουμε τις δημοκρατικές ανάγκες, τις, την ανάγκη διαφάνειας με παγκόσμια κλίμακα διεθνής αν θέλετε διαπραγματεύσεις. Θα πω μας το εξή και είναι προσωπική μου άποψη. Έχουμε παράδειγμα από την ε, εμπειρία του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή σε έναν άλλον τελείως διαφορετικό τομέα διαπραγμάτευσης τη μεταφορά δεδομένων, προσωπικών στοιχείων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο μηχανισμός που προέκρινε η Επιτροπή ξέχασε εντό εισαγωγικών τι ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δημοσιολογητή και άλλων. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς, εσείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό να μην επαναληφθεί. Δεύτερον, δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες όσον αφορά την διαπραγμάτευση, την τρέχουσα διαπραγμάτευση. Γιατί ανάφερα και στην δική μου εισήγηση ότι πρόκειται για μια αποσπασματική διαδικασία ανοργάνωτη με θύμα την διαφάνεια. Το κατά πόσον το αποτέλεσμα το απότοκο των διαπραγματεύσεων είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ε, είναι κάτι το οποίο θα γίνει το πολύ αργότερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα για κάποια τελικά σχόλια. Πρόεδρε, πιστεύω ότι μάθαμε πολλά σήμερα από πολλές διαφορετικές απόψεις και ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθηγητά ευχαριστώ πολύ που περάσετε αυτέ τι ώρε μαζί μα Να δώσω ένα παράδειγμα όμω πρώτα απ' όλα, γιατί αναφέρατε το ζήτημα τη βενσίνης. Ήταν ε, δικός μου φάκελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από πολύ καιρό, πάνω από 10 χρόνια πριν, και ξέρετε τι συνέβη. Είχαμε έναν μόνιμο διάλογο μεταξύ μέλων του Κογκρέσου και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάθαμε όμως ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καλύτερα εξοπλισμένη, αν θέλετε, πιο έτοιμη να μεταβάλει τα πρότυπά σε σχέση με ένα μόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικώς υιοθέτησε τα πρότυπα της Καλιφόρνιας για τα καύσιμα που ήταν τα καλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έγινε εν τέλει. Αφού όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε παίξει τον ρόλο του στην ε, διαδικασία, καθώς ήμασταν υπέρμαχοι της ποιότητας του αέρα. Πολύ αργότερα τα υψηλά αυτά πρότυπα εφαρμόστηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε διαφορετικοί, έρθανε κακήθεν του Ατλαντικού, όσον αφορά τους θεσμούς μας, τις αρμοδιότητες, τα διάφορα επίπεδα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μόνο και μόνο επειδή συζητούμε τώρα την TTIP τα πράγματα έχουν ξαφνικά βελτιωθεί ή απλουστευθεί. Ευχαριστώ και πάλι κύριε καθηγητά. Το σίγουρο είναι ότι τα θέματα αυτά είναι ενδιαφέροντα, σημαντικά, είναι πολιτικά, αφορούν την υγεία των ανθρώπων, τον εξυγχρονισμό διαφόρων τομέων τη βιομηχανία. Πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε έναν μηχανισμό λογοδοσίας κατέρθεν του Ατλαντικού άκουσα κάποια ενθαρρυντικά λόγια, αν δεν κάνω λάθο και να πω σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητή Goldman στην αρχή. Με την θέσπιση των πέντε αυτών αρχών, με την ενσωμάτωση των πέντε αρχών στι ευρωπαϊκέ διοικητικέ διαδικασίε. η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπνέει και ανέβει προ τα εμπρό και βελτιώνει τα πρότυπα σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και όταν θα μιλήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσθέσω αυτά στη σημειώση μου γιατί βλέπω εκεί κάποιον σκεπτικισμό, κάποιους δισταγμούς όσον αφορά τη θέσπιση βάση του άρθρου 298 της συνθήκης της Λισαβόνας των σχετικών διαδικασιών με βάση τα, τις αρχές που είπατε. Πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια ενοποιημένη νομοθεσία για την διοικητική διαδικασία θα ήταν καλή για την λογοδοσία μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι καλό για την διοίκηση, για τι διοικητικές διαδικασίε και θα επηρεάσει, ελπίζω, και το διεθνέ επίπεδο. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά ευχαριστώ πολύ πραγματικά που σήμερα μας δώσατε την ευκαιρία να ακούσουμε όλες αυτές τις ομιλίες. Στην Επιτροπή μας, σε αυτή την Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσει, οι διαβουλεύσει όσον αφορά την αξιολόγηση επιπτώσεων, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο που θα έχουμε πετύχει και διαφάνεια όσον αφορά τις διαβουλεύσει. Οι προτάσεις από την ομάδα δεν μας λένε και πολλά, δεν ε, είναι ικανοποιητικέ τελικώ. Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο μα. Να απλουστεύσουμε εν τέλει την νομοθεσία και να βελτιώσουμε την ποιότητά της χάρη σε ανάλυση επιπτώσεων, χάρη σε διαβουλεύσει. Είμαστε ακόμα μακριά από ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Πάντως, χάρηκα που άκουσα και με τον κύριο Χάρτεν ότι για αυτού του είδου τι διαβουλεύσει υπάρχουν κάποιες καλέ πρακτικέ μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Αναφέρεται την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη διαφάνεια και το τι έκαναν για τη διαφάνεια τελευταία, πω βελτίωσαν του κανόνε του. Καλό παράδειγμα. Και τέλο είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι τόνισε ο Πολωνός καθηγητής ο κ. Βιεζεμπόσκη. Διότι τις διοικητικές διαδικασίες στην Ευρώπη δεν τις αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ για τα παραδείγματα που μας δείχνουν πώς αναπτύχθηκε, πώς προχώρησε προς τα εμπρός η πολωνική διοικητική μηχανή. Έχω και εγώ στην Φιλανδία παραδείγματα μέχρι το 1809, άλλωστε ένα ε, μέλη, μέρος της Πολωνίας. Μετά γίναμε κομμάτι της Ρωσίας το 1809 και πρέπει να πω ότι έναντι της αυθαιρεσίας ο καλύτερος μηχανισμός αμυνάς μας ήταν το, οι διοικητικές διαδικασίες. Έτσι επιβιώσαμε και στην τσαρική Ρωσία. Γελάει εδώ ο Πολωνός Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε, δώσαμε τη μάχη κατά της αυθαιρεσίας, χάρη ακριβώς στις δικαιωτικές διαδικασίες. Έτσι επιβιώσαμε. Ο νόμος λοιπόν τα κατάφερε πολύ καλά και δεν επεξήλθε εναντί των εγώ των καταπιεστών. Αυτό το οποίο είπε λοιπόν ο κύριος ε, Χάντιν είναι ένας εξαιρετικός καταλόγος των λόγων για τους οποίους το Κοινοβούλιο πρέπει αμέσως να ξεκινήσει το σχετικό έργο για το διοικητικό δίκαιο Όντως, η συνθήκη το επιβάλλει, μεταξύ άλλων, πολλές φορές, ακόμα και η ίδια η Κομισιόν δεν το ερμηνεύει σωστά, ε, και λέει ότι ναι, είναι ένα ίσως, όχι, η, η συνθήκη το επιτάσσει. Επίσης, η συνεκτικότητα και συνάφεια των διοικητικών διαδικασιών και η νομιμοποίηση τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια έννοια που ανέφεραν πολλοί. Τελευταίο σχόλιο. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ για την TTIP, πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα ανώτερο επίπεδο διοικητικών διαδικασιών ακριβώς εν ώψη διεθνών διαπραγματεύσεων. Περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη αποτελεσματικότητα. Όλοι θα βγούμε καλύτεροι από αυτό, θα μάθουμε. Η πρόκληση είναι σημαντική. Όλοι στην Ευρώπη ανησυχούν για βάσιμους λόγους, ακριβώς λόγω της έλλειψης νομιμοποίησης, λογοδοσίας και του καθεξής. Κύριε Στιούαρτ, κύριε καθηγητά, έχετε δίκιο. Χρειάζεται περισσότερο διάλογος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά που περάσετε αυτέ τι ώρες μαζί μας. Ας συνεχίσουμε το διάλογο. Γνωρίζω ότι Δύο από εσά ε, ήταν μέλη και της ομάδας πανεπιστημιακών που συνέγραψε την πρόταση για νομίζω η κυρία Μέντες και ο κ. Βιεσμπόφσκι ήταν στην ομάδα ε, συζήτησης των ευρωπαϊκών διοικητικών διαδικασιών. Όλο αυτό θα κάνει καλύτερη την διακυβέρνηση και από αυτήν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Ε, may I thank all our distinguished speakers. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Εδώ και εκεί δεν είναι το Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ που συμμετάσχετε, που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτό κλείνει και η σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με το σημείο 25 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση από την κυρία Μαργκότ Φρέλιγκερ του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Κυρία Φρέλιγκερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με προσκαλέσατε. Προσλήθηκα να παρουσιάσω πώ έχει η κατάσταση εφαρμογή ε, ε, του ενιαίου ε, διπλώματο ευρεσιτεχνία όσον αφορά και το Διοικητικό Συμβούλιο και τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Συγγνώμη. Παρακαλώ, ο κύριος εδώ μπροστά να μην συνομιλεί με το διπλανό του. Εντάξει, συγγνώμη που σας διέκοψα. Εντάξει. Madame, please Μπορείτε να συνεχίσετε κυρία μου. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να επεξηγήσουμε το πώς έχει ο βαθμός ε, εφαρμογής ε, του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να εξετάζουμε πρώτον το νομικό πλαίσιο για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δεύτερον την προσέγγιση και έννοια του ενιαίου διπλώματος ε, ευρεσιτεχνίας που είναι πολύ συγκεκριμένη υπόθεση και τρίτον το συγκεκριμένο βαθμό ε, εφαρμογής που προβλέπεται από τον Ευρωπαίο Νομοθέτη για την εφαρμογή όλων αυτών. Αρχίζω, ξεκινώ με το νομοθετικό πλαίσιο. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δημιουργήθηκε από δύο κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2012 σχετικά αντίστοιχα αφορούν τη δημιουργία ενιαίων διαδικασιών και ενιαίας ε, προστασίας καθώς επίσης ε, και τις ε, συμφωνίες μεταφοράς και εκτέλεσης. Και τα δύο αυτά στοιχεία υιοθετήθηκαν με την διευρυμένη όπως αποκαλούμε συνεργασία Enhanced Cooperation που επελέγει ως ίστατη διαφυγή ε, προσφυγή όταν κατέστη σαφές ότι στο Συμβούλιο η απαιτούμενη ομοφωνία για τις διαδικασίες μετάφρασης ή μεταφοράς δεν μπορούσαν να επιτευχθούν όπως ήταν αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την διευρυμένη συνεργασία, enhanced cooperation, εκτός Ισπανίας και Ιταλίας που απέχουν για γλωσσικούς λόγους, αλλά επίσης και την Κροατία η οποία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έγκριση αυτών των κανονισμών όμως η Κροατία. Επιπρόσθετα η Ισπανία εισήγαγε μια προσφυγή για ακύρωση κατά αυτών των δύο κανονισμών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 10, Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για το οποίο θέμα ε, κατέθεσε τα συμπεράσματά του ο Γενικός Εισαγγελέας το Δεκέμβριο πέρυσι. Ε, συνέστησε να απορριφθούν αυτές οι προσφυγές. Όμως αναμένεται ακόμα η νομολογία, η απόφαση του δικαστηρίου κατά τους επόμενους μήνες. Αυτοί οι κανονισμοί ήδη άρχισαν να ισχύουν. Από την άλλη όμως πλευρά δεν εφαρμόζονται ακόμα, δεν είναι εφαρμόσιμοι ακόμα. Θα εφαρμοστούν μόνο από κοινού με την έναρξη σε ισχύ της συμφωνίας για το ενιαίο αυτό ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, UPC. Σε σχέση με το ενιαίο αυτό δίπλωμα ε, αφορά μια ε, διεθνή συμφωνία που στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα ενιαίο δικαστήριο ε, προσφυγής για θέματα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στις διαδικασίες της διευρυμένης συνεργασίας, Enhanced Cooperation. Εξαρτήθηκε από την έναρξη σε ισχύ η όλη αυτή εφαρμογή του ενιαίου δικαστηρίου ε, διπλωμάτων τεχνίας, ε, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οποιοδήποτε κίνδυνοι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Διότι φοβήθηκαν τα μέλη ότι χωρίς ένα ενιοποιημένο τέτοιο ε, όργανο προσφυγής η ενιαία, η ενιαία εφαρμογή θα αποτελούσε πρόβλημα θα ήταν προβληματική και θα υφίστατο ο κίνδυνος εθνικά δικαστήρια στα κράτη-μέλη με σχεδόν καθόλου ή πολύ μικρή εμπειρία και πείρα σε σχέση με θέματα επιδιαιτησίας ή εκδίκασης ε, θεμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να θέσει ένα αμφιβόλο την προσπάθεια αυτή των 25 κρατών μελών και θα δημιουργεί το μια μεγάλη νομική ανασφάλεια για τους χρήστες. Η συμφωνία για το ενιαίο αυτό δικαστικό σώμα ε, απαιτεί για την έναρξη σε ισχύ 13 επικυρώσεις ε, επιμέρους. Έξι κράτη-μέλη έχουν ήδη επικυρώσει. Περαιτέρω επικυρώσεις βρίσκονται καθοδόν. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι επικυρώσεις που απαιτούνται θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν διαδικαστικά κατά τα τέλη του 2015 εφέτος ή κατά τους πρώτους μήνες του 2016 και έτσι λοιπόν οι δυνατότητες ε, των ενιαίων αυτών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με βάση αυτό το ενιαίο όργανο δικαστικό θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Αλλά αναμένουμε ότι κατά τα μέσα του επομένου έτους ε, όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα. Επιστρέφω στην σύλληψη ή προσέγγιση ως ιδέα αυτού του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είναι ένα πιο σύνθετο θέμα και θέτει κάποιες δυσκολίες κατανόησης. Ε, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όπως αποκαλείται το ευρωπαϊκό δίπλωμα, ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας <clears throat> δεν έχει κάποιον αυτόνομο ξεχωριστό τίτλο είναι ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας υπό τους κανόνες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Και μόνο όταν έχει χορηγηθεί ένα τέτοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι δύο αυτοί οι κανονισμοί της ΕΕ μπορούν να εφαρμοστούν και να ισχύσουν. Όταν ένας ιδιοκτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει ε, λάβει αυτή την αναγνώριση από την υπηρεσία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τότε μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Και αν ζητήσει την καταχώρηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο ενιαίο Μητρό, αυτό θα σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα οι τρέχουσες διαδικασίες ε, της εθνικής κύρωσης ε, από τα διαφορετικά κράτη-μέλη επιμέρους θα υποκατασταθούν από μία κύρια διαπίστευση ή πιστοποίηση από πλευράς του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενιαία. Δεύτερον, η τρέχουσα αυτή τη στιγμή ρύθμιση για ε, τέλη ετήσια που πρέπει να καταβάλλονται, να πληρώνονται στις εθνικές αρχές για διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα αντικατασταθούν και θα υποκατασταθούν από ένα ενιαίο ε, τέλος το οποίο θα καταβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας. Και τρίτον, οι απαιτήσει όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή για μεταφράσεις σε πολλά κράτη-μέλη θα αρθούν, θα καταργηθούν και μόνο σε μια μεταβατική περίοδο κατά το μέγιστον 12 ετών θα υπάρξει μία ε, μετάφραση σε μία γλώσσα ε, ενωσιακή που θα απαιτείται ώστε η μετάφραση αυτή να υποβάλλεται σε, σχετικά, σε σχέση με σχετικά κείμενα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Είναι σημαντικό όμως να κατανοηθεί ότι αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υποκαταστήσει 100% πλήρως τις εθνικές ε, επικυρώσεις. Διότι αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα είναι μια πρόσθετη επιλογή για τους ε, ιδιοκτήτες κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Θα εξακολουθούν αυτοί να έχουν την δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να επικυρώνουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνία τους σε εθνικό επίπεδο κράτο, κράτος μέλος ή κράτη-μέλη αν αυτό επιθυμούν. Ε, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία θα είναι μια επιπρόσθετη επιλογή για ιδιοκτήτες, για κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από ένα τέτοιο δίπλωμα. Δεν θα υποκαταστήσει όμω όλες τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται εθνικά. Ο λόγος για αυτή την περίπλοκη σύνθεση ως ε, επικοδόμημα αυτού, αυτής της πρότασης για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα είναι πολυσχηδής η λόγη αυτή. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο νομοθέτης ήθελε ε, να εστόχευε, να οικοδομήσει στην προηγούμενη δομή σε σχέση με το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα όσον αφορούσαν ε, οι διατάξεις στα θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να υπάρξει ένα αξιόπιστο πλαίσιο στη συνέχεια μιας Ευρωπαϊκής Σύμβασης που θα διείπε τα θέματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έρχομαι τώρα στο επόμενο θέμα. Η δομή αυτού του Ευρωπαϊκού Διπλώματος με ενιαία δομή έχει φυσικά σημαντικές επιπτώσεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα εφαρμόζεται. Η διοικητική αντιμετώπιση του ενιαίου αυτού διπλώματος ευρεσιτεχνίας επομίστηκε και επιφορτίστηκε ως θέμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο. Ωστόσο δεν είναι κάποια αυτόνομη ξεχωριστή λειτουργία. Αυτή τη στιγμή εποπτεύεται και βρίσκεται υπό την, ε, τον, τον έλεγχο εποπτικά από τα κράτη-μέλη, από μια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε για αυτό το στόχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κυβερνών σώμα υπεύθυνο για τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και συντίθεται, συντίθεται, απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και από έναν επόπτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η επιλεκτική η, ε, η επιτροπή ε, η οποία υποπτεύει όχι μόνο αυτές τις δραστηριότητες αλλά έχει επίσης και τα καθήκοντα του να υιοθετεί τις ε, εκτελεστικές ε, ρυθμίσεις και διατάξεις που απαιτούνται για τις, ε, την εφαρμογή των όσων προβλέπονται για την έναρξη σε ισχύ του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και μέσα στις, πρωτο, στις δευτερογενείς εφαρμογές και ρυθμίσεις έχουμε ρυθμίσεις που αφορούν τις διοικητικές διαδικασίες και αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την Επιτροπή αυτή εποπτείας αλλά υπάρχει και η ανάγκη των τελών που πρέπει να καταβάλλονται όσον αφορά την ανανέωση τελών που θα καταβάλλονται ή πρέπει να καταβάλλονται από κατόχους ε, του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Και αυτό θα είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και να διεκπεραιώνει ε, η Επιτροπή Επιλογής ε, και Εποπτείας. Και ερχόμαστε τώρα στο άρθρο 12 του νέου κανονισμού που απαριθμεί ε, σχετικά κριτήρια που πρέπει να εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των τελών. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων είναι το μέγεθος της αγοράς, το επίπεδο τελών που αυτή τη στιγμή καταβάλλονται για ένα μέσου όρου, για ένα μέσου όρου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, αλλά επίσης και λήψη υπόψη συγκεκριμένων φορέων όπως πανεπιστημίων, ε, ιδρυμάτων έρευνας ε, και από την άλλη πλευρά έχουμε την ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που προβλέπει ως διάκταξη ότι το ανανεούμενο τέλος πρέπει από με τα διαδικαστικά τέλη διαδικασιών που πρέπει να καταβάλλονται στην υπηρεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για την εξέταση αιτήσεων Όλα αυτά από κοινού πρέπει να είναι επαρκής ε, όσον αφορά το άθροισμά τους, ώστε να υπάρχει ισοσκελισμός ε, όσον αφορά τα έσοδα ε, και τις δαπάνες, τον ισολογισμό δηλαδή του, της υπηρεσίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό διότι μέχρι σήμερα είχαμε ίσπραξη τελών ανανέωσης από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν τμήμα των εσόδων. Ένα τρίτο περίπου ε, των κονδυλίων σε σχέση με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας και πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της ε, χορήγησης ε, αδείας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας των προχορήγησης διαδικασιών. Αν είναι υπερβολικά χαμηλά αυτά τα τέλη, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αυξηθούν τα διαδικαστικά τέλη τα οποία θα έπρεπε να εισπράττονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνώρισε ο Ευρωπαίος νομοθέτης ως ζήτημα και έτσι επεθύμησε και θέλησε να αποφευθεί μια τέτοια κατάσταση ο νομοθέτης. Τι απορρέει, τι απορρέουν από όλα αυτά. Απορρέουν εν κατακλείδη, εν συντομία, ότι τα νέα τέλη πρέπει να είναι επαρκώς χαμηλά ώστε το ενιαίο αυτό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να είναι θελκτικό για τους χρήστες. Δεν μπορεί όμως να είναι υπερβολικά χαμηλό το επίπεδο αυτών των τελών, διότι δεν μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο η ισορροπία, ο ισοσκελισμός των εσόδων και των δαπανών της υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν με, τις, ε, με την αντίστοιχη ε, μονάδα για τα συμφέροντα των χρηστών και οι χρήστε ε, τοποθετήθηκαν και είπαν ότι δεν θέλουν να δαπανούν, να καταβάλουν περισσότερα για τα ανανεωμένα τέλη σε σχέση με τα όσα καταβάλουν σήμερα για παραδοσιακής μορφής διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία πιστοποιούνται και δια, ε, ε, την χάνουν διαπίστευσης από διαφορετικά κράτη-μέλη. Ως προς όλες αυτές τις ε, πτυχές ε, υπήρξαν στατιστικά στοιχεία τα οποία ε, συνελέγησαν και διετέθησαν στους χρήστες και στα κράτη-μέλη. Και αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σε κάποια κράτη-μέλη όπου υπάρχει τέτοια πιστοποίηση μειώνονται διαρκώς αυτά. Αυτή τη στιγμή κατά μέσον όρον πιστοποιείται ένα τέτοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε τέσσερα κράτη-μέλη από τα 25 που συνολικά σήμερα συμμετέχουν στη διαδικασία διευρυμένης συνεργασίας και 65% όλων των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πιστοποιούνται μόνο σε τρία κράτη-μέλη και σε λιγότερα από τρία κράτη-μέλη. Σαν συνέπεια όλων αυτών, οι χρήστε επιχειρηματολογούν και λέγουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν το επίπεδο τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται γι' αυτό θα είναι υψηλότερο από το επίπεδο των τελών που καταβάλουν σήμερα σε σχέση με την ανανέωση αυτών των διπλωμάτων σε σχέση με τα τρία ή τέσσερα κράτη-μέλη στα οποία διαπιστεύονται, ε, πιστοποιούνται αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας διακρατικά. Γιατί κάτι τέτοιο θα καθιστούσε, αν ήταν υψηλά τα τέλη, μη θελκτικό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία ανησυχούν ότι ένα χαμηλό επίπεδο εσόδων θα δημιουργούσε πολύ μικρότερα έσοδα για την ανανέωση, για την υπηρεσία, αλλά επίσης και για τα κράτη-μέλη για να ε, δοθεί το περιθώριο στα κράτη-μέλη να διεξαγάγουν ενημερωμένες πλήρως συζητήσεις ε, δόθηκαν στοιχεία χρηματοοικονομικά στα κράτη-μέλη και προβλέψεις, ε, προγνώσεις για το μέλλον ως προοπτικές ε, για το τι θα μπορούσε να συμβεί και τις επιπτώσεις όλων αυτών στο, στην χρηματοοικονομική ισορροπία των πραγμάτων για την υπηρεσία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχουμε 48 τέτοια πρότυπα τα οποία πιλωτικά εξετάστηκαν και συζητήθηκαν και οι συζητήσεις τι απεκάλυψαν απεκάλυψαν ότι ένα επίπεδο τελών το οποίο θα ανταποκρινόταν στο ισοδύναμο για ανανέωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε, σε τρία κράτη-μέλη σίγουρα θα ε, μπορούσε να συνεισφέρει στο να μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές ε, διαρροές εσόδων ένα επίπεδο τεσσάρων ή πέντε κρατών μελών αντίστοιχα σε σχέση με τα τέλη αυτά θα μπορούσε να θεωρηθεί εφικτό. Ένας άλλος ε, αριθμός στοιχείων που εξετάστηκαν από την Επιτροπή είναι το ζήτημα του αν θα έπρεπε να υπάρχει εξειδικευμένη ε, ειδική μείωση τελών για συγκεκριμένους φορείς συλλόγου ενώσεις όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα σε αυτό το σημείο οι απόψεις ε, των κρατών μελών και των χριστών συγκλίνουν περισσότερο, γιατί οι ενώσεις και σύλλογοι χριστών ε, έχουν επιφυλάξεις όσον αφορά μια τέτοια ε, μείωση ή έκπτωση τελών θεωρούν οι ενώσεις αυτές ότι είναι πιο σημαντικό να υπάρχει ένα γενικό επίπεδο τελών που θα είναι επαρκώς χαμηλό ώστε να είναι θελκτικό για, όλους ε, τους, ε, για όλα τα είδη και ομάδες κατηγορίες ε, χρηστών ή κατόχων και να υπάρχει ένας έλεγχος και αντιμετώπιση των, μέτρων, των κινδύνων να υπάρξει οποιαδήποτε κατάχρηση της κατάστασης με μείωση τελών. Λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη, η Υπηρεσία Διπλωμάτων ευρεσιτεχνία είναι έτοιμη τώρα να υποβάλει συγκεκριμένε, εξειδικευμένε προτάσεις για τη διαμόρφωση των τελών και στοχεύουμε στο να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των συντελεστών και παραμέτρων που αυτή τη στιγμή δημιουργούν κάποιε τριβέ ή προβλήματα. Ο στόχος ποιος είναι, να υποβληθούν προτάσεις και να κατατεθούν στην ε, Επιτροπή Επιλογής ε, για μια πρώτη συζήτηση κατά τα τέλη Μαρτίου 2015 με στόχο το επίπεδο τελών να, να εγκριθεί τον Ιούνιο. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εγκριθεί αρκετά νωρί το επίπεδο των τελών που θα ισχύει, ώστε να μπορέσουν να προσχεδιάσουν, να προγραμματίσουν τι ε, εργασίε του και να προσαρμοστούν στου αναγκαίου αυτούς υπολογισμού καταβολή τελών οι επιχειρήσει και οι επιχειρηματίες. Γνωρίζουμε τι δυσχέρειες που υφίστανται και τι δυσκολίε που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει επαρκή βούληση και θέληση από πλευρά κρατών μελών να υπάρξει μια συμφωνία επί επίπεδου τελών που θα διασφαλίζει ότι το ενιαίο αυτό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που περίμενε να ευδοκιμήσει και να μπορέσει να καρποφορήσει πάνω από τέσσερις δεκαετίες θα μπορέσει να προαχθεί επιτέλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την προλαλήσαντα προλαλήσασα για την ε, εξειδικευμένη περιεκτική παρουσίαση αυτών που συναποτελούν τα θέματα του ενιαίου ε, αυτού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κοινοβουλίου και του, ε, και του Συμβουλίου. Η ερώτησή μου επικεντρώνεται σε μια πολύ σημαντική πτυχή την διοργάνωση της ε, ε, ε, δικαιοδοσίας για τα δικαστικά σώματα ή τους φορείς που θα επιληφθούν αυτών των θεμάτων. Πώς έχει το πράγμα αυτή τη στιγμή. Το θέμα των περιφερειακών δικαστηρίων φαίνεται ότι έχει ήδη αποφασιστεί ή όχι. Ή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις επ' αυτού. Ευχαριστώ. Κύριος Λεμπρέτον. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα στην κυρία Φρόλιγκερ. Πρώτον, αν όντω αναμένουν τόσο πολύ τα κράτη-μέλη το ενιαίο αυτό δίπλωμα ευρεσιτεχνία, ισχύει αυτό στην πράξη, γιατί από ό,τι είδαμε υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία από τα κράτη-μέλη, υπάρχει όντω απαραίτητη πολιτική βούληση, πρώτο ερώτημα, δεύτερο ερώτημα. Η δυσπιστία αυτή των κρατών μελών μήπως τελικά οφείλεται σε άλλου λόγου, όχι αναγκαστικά οικονομικούς, δηλαδή ότι μπορεί να τεθούν εν κινδύνο, εν αμφιβόλωτα εθνικά διπλώματα βρεστεχνίας. Είπατε ότι το νέο αυτό δίπλωμα βρεστεχνίας θα συνεπάρχει με τα εθνικά διπλώματα βρεστεχνίας. Θεωρώ ότι στην πράξη θα είναι κάπως δύσκολο αυτό. μήπω τελικά αντιτεθεί, αντιταχθεί το ευρωπαϊκό αυτό δίπλωμα βρεστεχνίας στα γαλλικά, για παράδειγμα, αντίστοιχα διπλώματα. Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποβάλει ερωτήσει, Αν όχι, Ας ακούσουμε τις απαντήσεις από, τον από την κυρία Φρέλιγκερ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει στη συνέχεια το λόγο. Κυρία Φρέλιγκερ, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζιεύκα, αναφερθήκατε πολύ σωστά στο ερώτημα αυτό που αφορά την δημιουργία του ενιαίου δικαστηρίου για το δίπλωμα βρεστεχνίας. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα αυτό το δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το EPO, αποτελεί απλό παρατηρητή της προπαρασκευαστικής αυτής επιτροπής που έχει ως στόχο να θεσπίσει, να καταρτήσει το νέο δικαστήριο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Παρακολουθούμε πάντως εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία και όντω, σε πολλές υπομάδες γίνεται πολύ εντατική εργασία για τη δημιουργία του δικαστηρίου αυτού, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου, για τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, για τον ενιαίο κανονισμό που θα πρέπει να διέπει το ενιαίο αυτό δικαστήριο και το δίπλωμα βρεστεχνίας. Λαμβάνονται επίση αποφάσεις όσον αφορά το προσωπικό, όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης και τις συνθήκες αποδοχών των δικαστών, αποφάσεις που άπτονται του γενικότερου νομικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ενίο αυτοδικαστήριο, και επίσης λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά τον προπολογισμό του ενίου αυτοδικαστηρίου για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αν όμω θέλετε αυτή τη στιγμή πιο λεπτομερεί πληροφορίε, τότε μπορείτε να καλέσετε τον επικεφαλής της Προπαρασκευαστικής επιτροπή, ο οποίος θα μπορούσε να σας δώσει πολύ πιο λεπτομερεί πληροφορίε από ότι εγώ, εκπροσωπώντας το EPO. Όσον αφορά τώρα τις περιφερειακές, τα περιφερειακά τμήματα, έχει αγκριθεί η δημιουργία ενός περιφερειακού τμήματος μεταξύ της Σουηδίας και των τριών βαλτικών κρατών. Προβλέπονται όμω και περαιτέρω συζητήσεις, εκτιλήσονται μάλιστα οι συζητήσει αυτή τη στιγμή μεταξύ Τσεχίας και Σλοβακία όσον αφορά τη δημιουργία ενό περιφερειακού τέτοιου τμήματο, και ανάλογες συζητήσει λαμβάνουν χώρα μεταξύ τη Ουγγαρία, τη Σλοβενία και της Κροατίας, μολονότι η Κροατία δεν έχει ακόμα υπογράψει τη συμφωνία για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία και για το ενιαίο δικαστήριο. Και άλλα κράτη-μέλη έχουν πει ότι θέλουν να δημιουργήσουν τοπικά περιφερειακά τμήματα, Οι συζητήσεις πάντως αυτές θα ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια του 2015. Τώρα, όσον αφορά το, ζήτη, το ερώτημα του κυρίου Λεμπρετών, που έχει να κάνει με τη σχέση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς επίσης και το, τη σχέση που θα υπάρχει με το ενίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, Πολύ σωστά θίξατε το ζήτημα ότι το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν υφίσταται μόνο στο πλάι των παραδοσιακών διπλωμάτων βριστεχνίας, αλλά βρίσκεται και στο πλάι των εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική επίπτωση όσον αφορά τον αριθμό των εθνικών ετοιμάτων, των εθνικών μάλλον διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που θα προκύπτουν ή ενδεχομένω να μειωθούν εξαιτία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ξέρετε ότι ε, οι διαδικασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο μια πιο ταχεία διαδικασία. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοστίζει λιγότερο από ό,τι αν ακολουθηθεί η ευρωπαϊκή οδός. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνύπαρξη μεταξύ ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και ενιαίου διπλώματο ευρεσιτεχνία, καθώ επίση και η παράλληλη συνύπαρξη των εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνία δεν θα είναι καθόλου προβληματική. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για την ενημέρωση όσον αφορά τι προπαρασκευαστικέ εργασίε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών Ελπίζουμε θα να καταλήξουμε και να μην περάσουν χρόνια πριν εφαρμοστεί η δέσμη μέτρων. Αλλά δεν είναι εύκολο, είναι αρκετά πολύπλοκο. Εν πάση περιπτώσει, η ευκολότερη πρόσβαση στην κοινοτομία και στα εργαλεία κοινοτομία είναι προτεραιότητα κλειδί της ε, Επιτροπής Juncker. Ο κατακαιρματισμό στα διπλοπαταβέρες τεχνίας κοστίζει πολύ κάνει τη ζωή δύσκολη στις καινοτόμους εταιρείε. Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και στο πολιτικό επίπεδο τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε κάποια στιγμή και αυτό σημαίνει κυρώσεις και από τα υπόλοιπα 7 μέλη, κράτη-μέλη. Ε, περιμένουμε όμως και από εσά, διότι στο κράτη-μέλη που τα γνωρίζετε πολύ καλά μπορείτε να μας βοηθήσετε να περάσει το μήνυμα. Σας αλφάς που σα κύριε Δουλεύει στον τομέα και ξέρει πόση αξία έχει οι εταιρείε να μπορέσουν ε, τις ιδέες τους να τις κάνουν καινοτομία, να περάσουν στην αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να γίνει αυτό πρέπει η διαδικασία να είναι εύκολη και χωρίς κόστος αν γίνεται. Πιστεύουμε επίσης ότι έχει κρίσιμη σημασία. Το κόστος τα τέλη να είναι ελκυστικά για τις εταιρείε. Γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει δίπλωμα μόνο για μια χώρα, αλλά εξαρτάται από τη στρατηγική της κάθε επιχείρησης. Να έχουν όμως αυτή τη δυνατότητα να φροντίσουμε, παραλαμβάνω, αυτό έχει σημασία, το, το σύστημα τελικά να είναι ελκυστικό για τις επιχειρήσει. να είναι κάτι εύχριστο από τις επιχειρήσεις. Ε, η Κομισιόν, προκειμένου, έχει δεσμευθεί, υποστηρίξει την υπόθεση αυτή και θα συμμετάσχει με όλη την επιχειρηματολογία της και θα ταχθεί βεβαίω υπέρ κύρωση τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Αυτό θα μας επιτρέψει ελπίζω να δρομολογήσουμε και τη σχετική συμφωνία στην πράξη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ίσως να κλείσουμε και με αυτή την παρουσίαση και να ευχαριστήσω την κυρία Φρόγκερ για την εισήγησή της. Και τώρα. 31. Σημείο 31. Μεταρρύθμιση του δικαστηρίου. Ο λόγος εκ μέρους της Προεδρίας τον κύριο Καλνίτσι. Κύριε Καλίντς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Σφαμποντά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να λάβω μέρο σε αυτήν την συνάντηση και να σα πω που βρισκόμαστε με την μεταρρύθμιση του δικαστηρίου. Είμαι υπουργό του Υπουργείο Δικαιοσύνη και θα είμαι επικεφαλή τη ομάδα που διαπραγματεύεται αυτήν τη μεταρρύθμιση μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου τα επόμενα λεπτά να σα πω πού είμαστε και πού πηγαίνουμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σα ενημερώσω ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο το Συμβούλιο σημείωσε σημαντική πρόοδο. Η τον Δεκέμβριο, στι 11 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, κατέληξε καταρχήν συμφωνία Τα στοιχεία αυτής της ε, μεταρρύθμισης ήδη παρουσίασε ο Υπουργός μου, Υπουργός Δικαιοσύνης, την Επιτροπή σας στη Γιούρη, τον Ιανουάριο. Ε, να συνοψίσω τα βασικά αυτά στοιχεία, εκεί που κατέληξαν δηλαδή τα κράτη-μέλη. Πρώτον, θα αυξήσουμε το πλήθος των δικαστών σε 56 στο βασικό δικαστήριο τρία στάδια. Το Σεπτέμβριο θα προσθεθούν 12 δικαστές. Το 2016 θα προσθεθούν άλλοι 7 και θα διαλυθεί το ειδικό τμήμα για τους υπαλλήλους και το 2018 θα προσθεθούν άλλοι 9 δικαστές. Αυτές οι τρεις φάσεις θα ενσωματωθούν με νομικά δεσμευτικό τρόπο στο καταστατικό του δικαστηρίου. Αυτή είναι λοιπόν η κατεύθυνση. Όσον αφορά το κόστος, πιστεύουμε ότι η μεταρρύθμιση δεν θα είναι και τόσο δαπανηρή, αν λάβουμε υπόψη μας, με τις εξοικονομήσεις που θα πραγματοποιήσουμε το μεταξύ. Στις φάσεις 1 και 2, κάθε επιπλέον δικαστής θα έχει τρεις νομικής γραμματής, νομικούς γραμματείς. Δεν θα γίνουν όμως άλλες ε, προσλήψεις στην φάση 3. Από το 2019 το συνολικό κόστος λειτουργίας του δικαστηρίου θα είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνήσαμε ήδη ότι το δικαστήριο θα υποβάλει κατέτος στοιχεία οικονομικά για τη λειτουργία του και τις υποθέσεις που διεκπεραιώνει. Αν χρειαστεί θα διατυπώσουν περαιτέρω προτάσεις. Σε κάθε φάση της διεύρυνσης του Γενικού Δικαστηρίου θα γίνεται και εκτίμηση της κατάστασης. Θα γίνονται απαραίτητες του τροποποίησεις, εφόσον χρειαστεί, το οποίο δεν θα επηρεάσει το πλήθος των δικαστών, αλλά θα αφορά τις άλλες πτυχές της λειτουργίας και των δαπανών του δικαστηρίου. Γενικό Δικαστήριο θα αναθεωρήσει την εσωτερική του οργάνωση και τον εσωτερικό κανονισμό, θα υποβάλει δε τις απαραίτητες προτάσεις πριν τον Ιανουάριο του 2019. Η Προεδρία διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη για την μεταρρύθμιση αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι η καλή στιγμή να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε τις ε, πολύ αναμενόμενες λύσεις. Έτσι θα λειτουργήσει σωστά το Γενικό Δικαστήριο και πιστεύουμε ότι αυτό θα φρατώσει το μέσο πρόθεσμο όσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον. Το Συμβούλιο των Δικαιωρικών Συλλόγων τη Ευρώπη, που εκπροσωπεί ένα εκατομμύριο δικηγόρου, είναι υπέρ αυτή τη μεταρρύθμιση. Όλοι αυτοί ανησυχούν για τι καθυστερήσει που εμφανίζονται στο Γενικό Δικαστήριο. Την τελευταία εβδομάδα ενημερώσαμε και την Κορυπέρ για την συμφωνία και τη μεταρρύθμιση. Η Προεδρία από εδώ και πέρα θα συνεχίσει τι επίσημε επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα. Το Συμβούλιο προβλέψει περαιτέρω επαφέ για να συζητήσει τι τροπολογίε, τα σχέδια τροπολογιών στο πλαίσιο ενός τετραμερούς διαλόγου. Να σα ενημερώσω επίση ότι η Προεδρία υπέβαλε στους εκπροσώπους των των μελών την μέθοδο επιλογής των πρώτων 12 δικαστών για τα κρατη που θα υποβάλουν υποψηφιότητες. Εννοείται ότι το άρθρο 255 θα ισχύσει και πάλι, θα λειτουργήσει η επιτροπή του σχετικού άρθρου και θα γίνει ότι χρειάζεται μεταξύ για την λειτουργία του δικαστηρίου για τους διοικητικούς υπαλλήλους των ότι ήταν πριν να στο Γενικό Δικαστήριο. Η μέθοδος αυτή βρίσκει σύμφωνα τα κράτη-μέλη, έτσι κάπως θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από περίπου τέσσερα χρόνια εντατικών προσπαθειών επετεύχθη η συμφωνία είμαστε τουλάχιστον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα έτσι ώστε η πρώτη ομάδα νέων δικαστών να προσθεθεί από τον Σεπτέμβριο στους υφισταμένους. Παρακαλώ για τα σχόλιά σας. Η Προεδρία, κατά τα άλλα, όπως είπα, προσβλέπει σε επικοινωνικέ συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Συντομότερων Δυνατών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Μαρίνο Επίντο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά έχω μείνει άναυδος ακούγοντας αυτή την παρουσίαση. Και πραγματικά έχω μείνει άναυδος, διότι από μια χώρα που υπέστη αυστηρότατα μέτρα περικοπών και λιτότητας όπως την Πορτογαλία από την οποία προέρχομαι απαιτήθηκε από τη χώρα μου την Πορτογαλία να περικόψουμε δημόσιες δαπάνες και να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των δημοσίων κρατικών δαπανών. Κυρίως υπήρξε περικοπή δαπανών και ούτε καν λήφθη υπόψη η προοπτική αύξησης δαπανών. Αυτή η μεταρρύθμιση και τοποθέτηση του Συμβουλίου μας λέει τα εξής και ζητώ την προσοχή σας γι' αυτό το δικαστήριο πρότεινε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών σε 12, 12 ε, δικαστές ε, από το 2011 μέσα σε 4 χρόνια. Καθώς δεν υπήρξε συμφωνία από πλευράς ε, του Συμβουλίου για αυτό τον διορισμό των 12 αυτών δικαστών, στο Συμβούλιο από 28 μέλη 16 παρέμειναν εκτός. 16 παρέμειναν εκτός στο περιθώριο. Και αυτό για αυτή τη φάση που διήρκεσε τρία χρόνια. Δώδεκα λοιπόν αντί για 28. Και θεωρείτε ότι με αυτό λύθηκαν λέει τα προβλήματα. Είναι ωραίο όταν δεν υπάρχουν δισταγμοί και επιφυλάξεις να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να επιφορτίζονται και να επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι καταναλω... Ε, φορολογούμενοι. Αυτό λοιπόν ας είμαστε σοβαροί. Κάθε δικαστή ε, κοστίζει κατά μέσον όρων συγκεκριμένα κονδύλια διότι δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν να έχει τέτοιο μισθό ένας δικαστής. Ένα εκατομμύριο λοιπόν κοστίζει ο κάθε δικαστής. Αυτό έχει αναφερθεί σε έκθεση που συντάχθηκε. Κάθε κράτος μέλος λοιπόν για το Συμβούλιο ε, έχοντας ένα σύνολο 28 θα πρέπει λοιπόν να υπολογιστεί και το διπλάσιο, το αντίστοιχο κονδύλιο. Ειλικρινά βρίσκομαι στο Ευρωκοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής για πρώτη φορά, αλλά πιστεύω ότι μεγαλύτερο σεβασμός θα έπρεπε να υπάρχει σε σχέση με τους Ευρωβουλευτές για τους, ε, τα κονδύλια των φορολογουμένων μας ε, και την χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων. Πώς μπορεί να πετάμε από τα παράθυρα τέτοια κονδύλια όταν σε κράτη όπως την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα υπάρχουν σημαντικότατες περικοπές των δημόσιων δαπανών και μάλιστα σε δομικές δαπάνες, διαρθωτικές δαπάνες που απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής από πλευράς μου. Είναι αναγκαίο, απόλυτα αναγκαίο αυτό το μέτρο. Δηλαδή αυτό, όποιος ζητά δηλαδή και υποβάλλει μια τέτοια πρόταση πρέπει να το δούμε. Το 2007, το 2007 υπήρχαν τάσεις οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι 28 αυτοί ε, με 300 ή 400 ε, δίκες ετήσια που είχαν το 2014 είχαμε 700 τέτοιες περιπτώσεις ή 800 με άλλα λόγια αυτός είναι ο λόγος για αυτή την τάση, έτσι. Και έχουμε έλλειψη δικαστών κιόλας. Και έχουμε περισσότερες δίκες που πρέπει να διευθετηθούν και μεγαλύτερη διάρκεια κιόλα λόγω αυτών των προβλημάτων. Τι γίνεται λοιπόν με του δικαστέ, Πρέπει να διαρωτηθούμε τι γίνεται με του δικαστέ και πώ λειτουργεί έτσι αυτή η πρωτοβουλία. Η επιχείρηση, μια επιχείρηση είναι το προϊόν των ε, ε, δράσεων των εργαζομένων εμείς πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ιδιαίτερα απαιτητικοί για την ανταγωνιστικότητα. Ποιος είναι ο αριθμός ε, ε, δικών που μπορεί ο κάθε δικαστής να αντιμετωπίσει. Ο δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη δική μου χώρα πολλές θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες δίκες. Αποφασίζουν στο πρωτοδικείο 300 ή 400 τέτοιες δίκες ή υποθέσεις οι δικαστές. 150 ε, τέτοιες δίκες επιλαμβάνονται ε, στο δευτερογενές. Στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε 90.000 περίπου υποθέσεις για 47 δικαστές. Στο Γενικό Δικαστήριο ο αριθμός που θέλουμε τώρα να διπλασιαστεί, ο αριθμός των δικαστών, έχουν 27 δίκες των οποίων υποθέσεις που επιλαμβάνονται έτος όλες και όλες. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο και δεν μπορούν να ξεπεράσουν και να αντιμετωπίσουν 40 ή 50 τέτοιες υποθέσεις να διευθετούν αιτήσια. Λοιπόν, αυτό το μέτρο, μια και έρχονται εδώ και το λένε αυτό, δηλαδή ζητεί το διπλασιασμό ε, σε σχέση με τα μέλη του το ε, δικαστήριο, νομίζω είναι μια προσβολή της ίδιας της νοημοσύνης των πολιτών ε, και σε σχέση με μένα το αναφέρω αυτό ως Ευρωβουλευτής που εξελέγει για να επα επαγρυπνώ σε σχέση με τις δαπάνες και να, με κριτικό πνεύμα να παρακολουθώ τα όσα γίνονται και βλέπω ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Γίνονται τέτοιες δαπάνες. Θα πρέπει να προστατευτούν οι φορολογούμενοι έναντι τέτοιων ε, μέτρων και της επιβολής ε, φόρων ταυτόχρονα από αυτούς τους ίδιους. Είναι αναγκαίο λοιπόν να θεσπιστούν αντικειμενικά στοιχεία παραγωγικότητας για τα δικαστήρια. Πρέπει να ξέρουμε το βαθμό αποτελεσματικότητας κάθε σώματος. Τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα μόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υφίστανται σε αυτή την, ε, τον έλεγχο αυτών αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας και δεν ξέρω πόσα κερδίζει ένας ε, δικαστής ε, ε, και που ο μισθός του μπορεί να είναι πολύ υψηλός. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την γενική του σταδιοδρομία που ξεπερνά κάθε πλαίσιο. Μπορεί να συμμετέχει και σε διάφορα συνέδρια, διάφορα σεμινάρια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και εφιστώ την προσοχή σε αυτά τα θέματα ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια μέτρα χωρίς να υιοθετείται η αρχή, το κριτήριο της παραγωγής ο αριθμός των δικών δηλαδή των υποθέσεων που πρέπει ένας δικαστής να μπορεί να διεκπεραιώνει ετήσια. Λοιπόν, ή εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των φορολογουμένων ή κάθε ένα κάνει ό,τι θέλει, δαπανά χρήματα, λέμε Α, δεν είναι δικά μα τα χρήματα, είναι ξένα χρήματα, α τα δαπανίσουν οι άλλοι όπω θέλουν. Λοιπόν, θα πρέπει να υποβληθούν αυτά τα θέματα σε αυτά τα κριτήρια. Να μην υπάρχει καμιά απόφαση για αυτά τα θέματα, εφόσον δεν θα έχουμε συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, τι πραγματικέ ανάγκε που υπάρχουν. <clears throat> Διότι υπάρχουν κριτήρια και καταστάσεις που είναι πολύ ανησυχητικές. Τώρα, <clears throat> σε σχέση για παράδειγμα με το πρωτοδικείο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστήθηκε, προτάθηκε να υπάρξουν αυτές οι δαπάνες. Θα είναι τώρα πολύ ακριβότερη η, ο διπλασιασμός ε, των ε, δικαστών ή το να έχουμε και την, ε, το δικαστήριο το οποίο θα συσταθεί για θέματα διπλωμα, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να στοχαστούμε και να προβληματιστούμε νυφάλια και ήρεμα και να μην πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Απαιτούμε αντικειμενικά αξιόπιστα στοιχεία για το κόστος, για την πραγματική κατάσταση, την παραγωγικότητα και ε, την αποτελεσματικότητα των δικαστών κάθε ε, σώματος και κάθε φορέα. Διότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει ε, σεβασμός στους λαούς, στους πολίτες της Ευρώπης που εμείς εδώ εκπροσωπούμε ως αιρετή εκπροσωπή τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέντε, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον όλο χρόνο που απαιτείται για τη διεκπαιρέωση μια δίκη στο δικαστήριο και αυτό επηρεάζει τελικά την οικονομία. Δηλαδή, αν η διεκπαιρέωση μια δίκη απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο χρόνο και αυτό αποτελεί τελικά πρόβλημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξετάζουμε το κόστο των επιπλέον δικαστών χωρί να λαμβάνουμε υπόψη μα τον χρόνο που απαιτείται για την εκδίκαση μια υπόθεση. Στόχο μα είναι η δικαστική διαδικασία να είναι γρήγορη, και αποτελεσματική. Μα απασχολούν λοιπόν οι ανησυχίε που εκφράσατε, αλλά από την άλλη θέλουμε να επιτελείτε σωστά και το δικαστικό έργο. Βασικό μα μέλημα θα πρέπει να είναι να έχουμε τον απαραίτητο αριθμό δικαστών προκειμένου να λαμβάνουμε αποφάσει ε, με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση τη εξέτασή μα. και αν υπερβούμε επίση και την αρχή του ένας δικαστής αναχώρα, όπως γίνεται προκειμένο, μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε και άλλα μελήματά μας, όπως το να έχουμε μια ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, να καλύψουμε διάφορους νομικούς τομείς. Σας ευχαριστούμε κύριο Ζεύκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου για όλες τις πληροφορίες. Ευθύς εξ αρχής στην παρέμβασή μου θέλω να παρακαλέσω ή δυνατόν εσείς να μας πείτε κάτι παραπάνω, να μας πείτε δύο λόγια για την μέθοδο της επιλογής των πρόσθετων αυτών δικαστών που από τα κράτη-μέλη θετικά αξιολογούν ή αξιολογήθηκαν, διότι αυτό το, αυτό το στοιχείο είναι πράγματι σημαντικό. Για την κυρία Ρέντα, ουσιαστικά ανέφερε τα περισσότερα αυτών που θα ήθελα εγώ να αναφέρω στη δική μου παρέμβαση. Μια και ο Πορτογάλος συνάδελφός μας τόσο συναισθηματικά φορτισμένο λόγο ε, εκφώνησε. Το θέμα αυτών των ε, ε, δράσεων είναι ένα θέμα το οποίο σε ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν πρόκειται μόνο για την αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου, αλλά για την ίδια την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι ο χρόνος, η συνιστόσα η χρονική που απαιτείται ώστε μία υπόθεση να διευθετηθεί από το δικαστήριο όλο και περισσότερο διαρκεί, γίνεται όλο και περισσότερο χρονοβόρα και περισσότερο κοστοβόρα. Λοιπόν, αυτό και αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβαρύνεται ιδιαίτερα. Όλο και μεγαλύτερα τέλη και ε, έξοδα απαιτείται να καλυφθούν. Διότι αυτό συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων για την λήψη αποφάσεων μέσα σε αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Έτσι λοιπόν μια επιχείρηση μπορεί μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα να χρεοκοπήσει, να πτωχεύσει. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί, να αλλάξει αυτή η κατάσταση πραγμάτων, ώστε να μπορεί να λειτουργεί κατά το βέλτιστο τρόπο το δικαστήριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα θα ήμουν ικανοποιημένος μπορώ να πω αν ο αριθμός των δικαστών διπλασιαζόταν. Και αν κάθε κράτος μέλος δεν θα είχε ένα, αλλά ίσως και δύο δικαστές. Αλλά τι βλέπουμε, εξοικονομήσεις, περικοπές. Αν πρέπει να περικοπούν κονδύλια και να γίνουν οικονομίες ε, και για το δικαστήριο, τι θα γίνει με τους 12 δικαστές. Η μεταρρύθμιση πρέπει να ολοκληρωθεί λοιπόν πλήρως συμπεριλαμβανομένου και του δικαστηρίου για τους ε, υπαλλήλους ε, η μεταρρύθμιση εκείνο που θέλουμε είναι να μην πολλαπλασιαστεί όσον αφορά τα έξοδά της. Να μην υπάρχει ανησυχία, δεν μπορεί να δράσει εκτός ελέγχου το δικαστήριο. Είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει λοιπόν τις δραστηριότητες του δικαστηρίου. Να γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ποια είναι τα κόστη γνωρίζουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να ρωτήσουμε και να διερωτηθούμε αν δεν μπορεί ή μπορεί ένας δικαστής να διευθετήσει 100 ή παραπάνω υποθέσεις ή όχι. Υπάρχουν όμως σημαντικά θέματα. Αν τα αντιμετωπίσουμε με ένα στενό πνεύμα θα είμαστε κατά της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Χαίρομαι όταν ακούω για την πρόοδο διότι η πρόοδος επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να προαθεί και δεν προαγόταν. Είχαμε τη γνωμοδότησή μας που είχαμε ετοιμάσει, το Συμβούλιο όμως δεν προχώρησε. Όταν λέει τώρα το Συμβούλιο ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να ληφθεί μια απόφαση μέχρι τις θερινές διακοπές ε, του 2015, ε τότε καλό είναι, τότε είναι πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, ας δούμε τι μπορεί να γίνει και αν είναι δυνατόν θα θέλαμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Mr. Le Breton. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεμπρετών έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ο κύριος Μαρίνο Επίντο, ο συναδελφός μου, με κάλυψε. Και εγώ με κατά του σχεδίου αυτού του διπλασιασμού του αριθμού των δικαστών. Πρώτον, θα κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Έχουν γίνει μάλιστα μελέτες. Κάθε δικαστής κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ ανά έτος. Επομένως, ε, καταλαβαίνετε ότι ε, θα κοστίσει η, το νέο αυτό σχέδιο επιπλέον 28 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Μας λέει ότι δεν πρόκειται να προσλάβετε επιπλέον προσωπικό, γραμματής κτλ. Είμαι σίγουρος θα προσλάβετε επιπλέον διερμηνείς για παράδειγμα, μεταφραστές και πολύ φοβάμαι επίσης ότι δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο αυτό δικαστήριο με τα επιπλέον αυτά μέλη. Θα αυξηθεί τελικά ο αριθμός των υποθέσεων, ναι, αλλά θα δοθεί προτεραιότητα κυρίως στις οικονομικές διαφορές. Επίσης, το άρθρο 257 του, της Συνθήκης της Λισαβόνας λέγεται ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να συστήσουν εξειδικευμένα δικαστήρια, εφόσον λέγεται λοιπόν αυτό από τη Συνθήκη, δεν λέγεται όμως αν μπορούμε να καταργήσουμε εμεί ένα δικαστήριο, όπω το Δικαστήριο Δημόσια Διοίκηση. Ένα ακόμα πρόβλημα, λίγο πιο προσωπική φύση, αν θέλετε, έχει να κάνει με το κόμμα μου, το Front και άλλα ανάλογα κόμματα. Το να διπλασιάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τους δικαστές ουσιαστικά σημαίνει ότι τους δίνουμε κίνητρο να επεμβαίνουν περισσότερο στην εθνική κυριαρχία. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω εγώ να αυξηθούν οι καταχρήσεις που ήδη είχαμε πάρα πολύ στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε και να περισσώσουμε το δικαστήριο, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη λύση που πρότεινε ο Μαρίνο Επίντο. Να βρούμε δηλαδή τρόπο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του δικαστηρίου. Είναι, θα πρέπει ίσως να εργαστούν λίγο περισσότερο δικαστές, δεν θα τους κάνει κακό. Τα όσα είπε ο κύριος Πίντο μπορώ να τα ακολουθήσω και να συμφωνήσω. Μια και με κριτικό πνεύμα τοποθετήθηκε κατά της πολιτικής λιτότητας και περικοπών του παρελθόντος και έναντι της Πορτογαλίας της ίδιας. Όμως η συγκρουσιακή αυτή σχέση δεν είναι σωστή νομίζω. Δηλαδή πολιτική λιτότητας έναντι διασφάλισης του κράτους δικαίου. Όταν ασκούνται τέτοιε επικρίσει, αυτέ πρέπει να γίνονται σε ένα άλλο πεδίο και όχι σε αυτό. Θέλω το αντίθετο να τονίσω ότι με την αύξηση των υποθέσεων και δικών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημιουργείται σήμερα μια κατάσταση στην οποία οι αποφάσει όσον αφορά τέτοιε υποθέσει απαιτούν ένα όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ω συνιστόσα χρονική. Μέχρι και 44 μήνες διαρκεί νομίζω η διαδικασία μέχρι να υπάρξει απόφαση που ε, θα ε, εκφράσει το δικαστήριο. Και όταν Έχουμε λοιπόν σε ένα κράτος δικαίου μια κατάσταση που πρέπει σε ένα εύθετο εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνονται τέτοιες διαδικασίες. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα, σήμερα. Και είναι σωστό αυτό το οποίο συζητήσαμε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και συζητήσαμε και στην επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τους ίδιους τους δικαστές. Είναι σωστό να καταλήξουμε σε μια διεύρυνση του αριθμού των δικαστών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες. Όταν διευρύνουμε, επεκτείνουμε τον αριθμό των δικαστών, μια ποσόστοση πρέπει να ε, προσδιοριστεί. Αν υποβάλλονται δύο προτάσεις από κάθε κράτος, ένας άνδρας, μία γυναίκα πρέπει να διορίζονται, ώστε η πρόθεση της ισότητας των φίλων να διασφαλιστεί και αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Πολλά προαναφέρθηκαν. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα πράγμα. Ένα πράγμα είναι σαφές. Έχουμε πραγματικά ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο, μια μεγάλη χρονική συνιστόσα, μεγάλη χρονική περίοδος απαιτείται για την διεκπαιρέωση τέτοιων υποθέσεων και μπορεί μια επιχείρηση να πτωχεύσει για παράδειγμα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δυνατόν παθητικά ως παρατηρητές ε, να παρακολουθούμε και να σταυρώνουμε τα χέρια. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν μεγάλες ε, δαπάνες και πρέπει να τεθούν προτεραιότητες. Εγώ πιστεύω η καλύτερη επένδυση είναι στον τομέα της δικαιοσύνης. Η καλύτερη επένδυση που μπορεί να επιτευχθεί όταν πρόκειται για την παραβίαση ή παράβαση κάποιου δικαιώματος στην Ευρωπολίτες προσφεύγουν, προστέχουν στη δικαιοσύνη. Όποιος καθυστερεί λοιπόν αυτό σημαίνει αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα. Λοιπόν, πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα με, με άλλα λόγια 20, 28 οσιδήποτε βουλευτές να υπάρξει επαρκής αριθμός. Όταν λέμε όμως 28 και δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια για την επιλογή τους, τι, κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την παραγωγικότητα αυτών των δικαστών. Ακριβώς όπως και με μια μηχανή για παράδειγμα. Ωραία, δεν είναι δυνατόν ε, ένας δικαστής με τον ίδιο τρόπο να εργάζεται. Εντάξει, είναι όμως σημαντικό ο αριθμός των υποθέσεων να είναι ε, αποτελεσματικός σε σχέση με τον αριθμό των δικαστών. Να δούμε τι γίνεται με τις δαπάνες για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ίσως θα πρέπει μισθοί βουλευτών ή κάποιων άλλων να περικοπούν για να υπάρξουν χρήματα να γίνουν οι επενδύσεις που ε, απαιτούνται στη δικαιοσύνη. Να είμαστε ταχείς, ε, να μπορούμε δηλαδή με ταχύτερους ρυθμούς να διεκπαιρεώνουμε υποθέσεις δικαστικά. Ευχαριστώ. Um, uh, Έχω δύο ερωτήσεις προς την Προεδρία. Όμως προηγουμένως επειδή πιέζει ο χρόνος και αφού κλείσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό έχουμε ένα σημείο το 27 που μας απομένει. Α, όχι, με συγχωρείτε λέει ο Πρόεδρος, το 26 είναι. 26 και 27 ε, θα τα κάνουμε απόψε. Τα υπόλοιπα αναγκαστικώ αναβάλλονται. Αυτό είναι μια ανακοίνωση, ενημέρωση για όσου ενδεχομένω περιμένουν εδώ στην αίθουσα για να ακούσουν κάτι για τα επόμενα σημεία. Δύο λοιπόν ερωτήσει προ την Προεδρία. Πρώτον, κατάλαβα καλά ότι στο, στην τρίτη φάση μεταρρύθμιση δεν θα δοθεί διοικητική βοήθεια στους τελευταίους νέους δικαστές. Και το παράδειγμα ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι αυτή η βοήθεια για την παραγωγικότητα του δικαστηρίου. Αυτό το βρίσκω λίγο προβληματικό. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο γενικό. Στην συνθήκη της νίκης τα κράτη-μέλη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λύση για το μέλλον είναι να δημιουργήσουμε ειδικευμένα σώματα και ξαφνικά τώρα πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ουσιαστικά καταργούμε ας πούμε το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρωτώ τα κράτη-μέλη το σκέφτηκαν σοβαρά αυτό. Γιατί αντιστρέφουν λοιπόν το άρθρο 256 αν δεν κάνω λάθος που προέβλεπε ακριβώς το αντίθετο και το οποίο περιλαμβανόταν στη συνθήκη της νίκης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Κύριε Σπόπολε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Η Προτρία σημειώνει όλες τις απόψεις και ερωτήσεις. Η βασική σας παρατήρηση είναι με βάση ποια στοιχεία προχωρούμε στην αύξηση του πλήθους των δικαστών. Λοιπόν, καταρχήν αναμένουν αυτή τη στιγμή αιτήματα αποζημιώσεων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν παγώσει εκατομμύρια ευρώ που εξαρτώνται από αποφάσεις του δικαστηρίου. Το σύστημα δεν λειτουργεί, τέλο πάντων δεν έχει τα καλύτερά του. Υπάρχει τεράστιος φόρτος λοιπόν ακριβών υποθέσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Η αύξηση του πλήθους των δικαστών είναι σαφώ μια λύση. Τώρα, χρειαζόμαστε 8. Ε, κοιτάξτε, η απόφαση αυτή είναι αναγκαστικά εν μέρη πολιτική. Τα κράτη-μέλη, αν με έναν ε, μικρότερο αριθμό, θα δυσκολεύονταν να καταλήξουν κάπου. Δεν θα καταλήγαμε ποτέ στη συμφωνία στο Συμβούλιο. Γι' αυτό και η λύση που προκρίνουμε είναι κάθε χώρα να πάρει ένα δικαστή και κάποια στιγμή το σύστημα θα ισορροπήσει. Να συζητήσουμε πάντως, αν θέλετε, τι ανησυχίες και του κυρίου Πίντο και του κυρίου Λεμπρετό. Να σας δώσουμε, αν θέλετε, περισσότερες πληροφορίες, ό,τι χρειάζεται. Είναι στη διάθεσή σας για να καταλάβετε που βασίσαμε τις αποφάσει μας. Κυρία Ρέντνερ και κύριε έχουν δίκιο. Ότι δηλαδή χάνουμε λίγο σε συνοχή. Και, και Σβιέσκα είπε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Η βασική αρχή κοιτάξτε είναι ότι θα έχουμε ένα καταλόγο κρατών μελών που θα ακολουθεί την εκπεριτροπής προεδρία με τη σειρά δηλαδή έτσι όπως η Γερμανία, μετά η Φιλανδία, μετά η Κροατία και ούτω καθεξής. Θα υπάρχει λοιπόν μια κλήρωση με την οποία θα καταλήξουμε σε ποια είναι τα, πρώτα 12 κράτη-μέλη με τα οποία θα ξεκινήσουμε. Θα φροντίσουμε επίσης την ισότιμη γεωγραφική κατανομή. Αυτή είναι η βασική αρχή. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτή είναι η μέθοδος. Και τα κρατη είπαν ναι για αυτήν την λύση. Για τις ερωτήσει του κ. Βόμποντα τώρα αφορούν ε, την ουσία του πράγματος, όντως. Και την τρίτη φάση, ναι, όντως, δεν θα δώσουμε επιπλέον γραμματική υποστήριξη, το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει μια εσωτερική μεταρρύθμιση, δηλαδή θα αναλογούν σε κάθε δικαστή 2, κάτι βοηθή Αυτό θα επηρεάσει κατά τη βεβαίωση τη δουλειά των δικαστών. Πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Δεν τώρα αν η κυρία θέλει να πει λίγο περισσότερα για το πώς θα επηρεαστεί το έργο των δικαστών και όσον αφορά τη συνθήκη της νίκαιας και το άρθρο 256 σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια ναι, ήταν μια ιδέα όμως το δικαστήριο στην πρότασή του έκρινε ότι η αύξηση του πλήθους των δικαστών και όχι τα ειδικευμένα δικαστηρία είναι η καλύτερη λύση για τα σημερινά προβλήματα. Και πάλι δεν ξέρω αν ε, η συνέντευξη μου θέλει να προσθέσει κάτι, αλλά αυτά είχα να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. okay, ε, ε, Μα... Μάλιστα λοιπόν μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο, επί του παρόντος τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Πρόεδρε, για μία προσαφήνιση σε σχέση με τον συνάδελφο για τον συναισθηματικά φορτισμένο τόνο της παρέμβασής μου. Εγώ δεν έχω κοινοβουλευτική πείρα, ούτε πολιτική πείρα και γι' αυτό τον λόγο, όταν κάνω λόγο και μιλάω για πράγματα που πιστεύω σε αυτά, μιλάω με την καρδιά μου και μιλάω συναισθηματικά φορτισμένα έτσι. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως έλεγα μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 26 παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την γνωμοδότηση παριθμών 2 κάθος 13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο στην νομική υπηρεσία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την σημαντική αυτή γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση παριθμών 2 κάθος 13 της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι υπάρχει ασυμβατότητα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σχέδιο προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως έτυχε διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο. Και ουσιαστικά η γνωμοδότηση αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Το δικαστήριο αποφάσισε να συνεδριάσει σε τμήμα μέγιστης σύνθεσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έδωσε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στην απόφαση αυτή. Πρωτού σας παραθέσω τώρα τους λόγους που διέπουν τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα ήθελα να σας δώσω λίγο το νομικό, αλλά και το νομικό πλαίσιο και να κάνω και μια σύντομη ιστορική αναδρομή της όλης υπόθεσης. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υπόθεση που στο παρελθόν δεν είχε απασχολήσει το δικαστήριο και για την οποία γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το δικαστήριο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού εξετάσει τα διάφορα αστικά επιχειρήματα έκανε πολύ σημαντικές προκαταρκτικές αναλύσεις. Είναι γνωστό επίση ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα τελευταία 45 χρόνια με δική της πρωτοβουλία δημιούργησε ένα κοινοτικό πλαίσιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων λαμβάνοντα κυρίως υπόψη την ιδιαιτερότητα του ενωσιακού δικαίου και εμπνεόμενο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και βασιζόμενο επίση στην ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Παράλληλα, η ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται πολύ από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία όλα τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη. Και μπορούμε να πούμε ότι ε, η σύμβαση αυτή υπερβαίνει ακόμα και τις συνθήκες της Λισαβόνας. Θα μπορούσαμε να περθούμε στην απόφαση της 13 Σεπτεμβρίου 1979, την υπόθεση Χάουερ, στην οποία το δικαστήριο αναφερόταν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρώντας ότι αποτελεί η σύμβαση αυτή πολύ σημαντικό μέσο προκειμένου να επιληθούν σχετικές υποθέσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την εποχή εκείνη ήταν το μόνο νομικό μέσο που υπήρχε για τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης το δικαστήριο έκανε μια, προχώρησε κοινή δήλωση με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωση του 1977 στην οποία αναφέρεται στην πρωταρχική σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι η ε, έμεση αυτή προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσε όχι μόνο να ενισχύσει αλλά να εμπλουτίσει περισσότερο την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έμεση όμως αυτή προσχώρηση θεώρησε ότι δεν ήταν επαρκή. Το 1990 λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα ανακοίνωση Επίσης το 1993 το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό και ήθελε ουσιαστικά να δει αν από νομικής πλευράς μπορεί να προσφορήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή του δικαστηρίου δεν είναι το πρώτο κείμενο το οποίο ασχολείται με μια ενδεχόμενη προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στη γνωμοδότηση 2 94 της, του Μαρτίου 1996 το δικαστήριο μετά από παρότρινση του Συμβουλίου είχε ήδη εξετάσει το αν ήταν σκόπιμη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθεαυτήν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τότε το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι δεδομένων των συνθήκων που ίσχυαν τότε, μία τέτοια προσχώρηση, η οποία κατά το δικαστήριο λάμβανε συνταγματικό χαρακτήρα δεν ήταν δυνατή εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένη νομικής βάσης και επομένως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσχώρηση μετά από τροποποίηση μόνο των συνθήκων. Η τροποποίηση αυτή όντως έλαβε χώρα από τότε που είχαμε δηλαδή την πρώτη αυτή γνωμοδότηση και μέχρι την γνωμοδότηση την τελευταία του Δεκεμβρίου 2014. Εφόσον στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το εξής πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως προς αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η διάταξη αυτή δεν αποτελεί εναλλακτική λύση, αλλά αποτελεί πλέον υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρέωση προσχώρηση λοιπόν και αυτό ακριβώς τόνισε και στο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν το Μάιο του 2010 αποφάθηκε για τη συνταγματική πτυχή της προσχώρησης Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη νέα αυτή νομική κατάσταση ζητώντας από το Συμβούλιο εντολή διαπραγμάτευσης και το Συμβούλιο έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2010 αυτή την εντολή διαπραγμάτευσης. Έκτοτε χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια μέχρι να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης το οποίο οριστικοποιήθηκε με συμμετοχή των θεσμικών οργάνων αφενός και, με τη συμμετοχή των αρμοδίων οργάνων από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφετέρου. Η συμφωνία αυτή δεν προέβλεπε απλώς και μόνο την προσχώρηση αυτή καθεαυτήν, αλλά προσπαθούσε επίσης να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες, τις θεσμικές και νομικές ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την αρμοδιότητα και το ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς αυτό λοιπόν το σχέδιο συμφωνίας προέβλεπε την πρώτερη εφαρμογή, εμπλοκή μάλλον, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα και εφόσον το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν είχε ήδη αποφανθεί για τα ζητήματα αυτά. Θεωρήθηκε λοιπόν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ότι θα μπορούσε να προχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο και στις 5 Μαΐου του 2010 το Δικαστήριο ήδη υιοθέτησε ένα έγγραφο περισυλλογής σε σχέση με την ενδεχόμενη προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, μέσω αυτού του σχεδίου συμφωνίας θελήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσε να συμμετέχει περισσότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Πώς θα γινόταν δηλαδή η εκλογή των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακολουθήθηκε λοιπόν η διαδικασία υποβολή γνωμοδοτήσεων και έτσι καταλήξαμε στη γνωμοδότηση 2 13 προκειμένου στα πλαίσια γνωμοδότησης αυτή να δούμε ποια ήταν η δυνατότητα συμβατότητα με τις συνθηκες Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωσης. Πολλά κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα υπέβαλαν κάποιε παρατηρήσει. Ποια είναι η επιχειρηματολογία που ακολούθησε το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Το Δικαστήριο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε εδώ πέρα μία εντελώς ε, διαφορετική προσέγγιση από αυτή που είχαμε στη γνωμοδότηση του 1996. Αναγνωρίζει ότι έχουν εξελιχθεί και τροποποιηθεί οι συνθήκες αφενός και αφετέρου πλέον το δικαστήριο είχε στα χέρια του ένα συγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας το οποίο υποβλήθηκε από τα θεσμικά όργανα. Το δικαστήριο λοιπόν αρχικά αναφέρεται στην σημαντική εξέλιξη του νομικού πλαισίου. Επιβεβαιώνει το δικαστήριο ότι οι φυστάμενες συνθήκες περιέχουν πλέον την κατάλληλη νομική βάση για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μολονότι δεν γίνεται σαφής αναφορά σε μια τέτοια υποχρέωση. Το δικαστήριο επίσης λέει ότι η προσχώρηση αυτή θα μπορούσε να γίνει χωρίς, μάλλον, θα μπορούσε να γίνει μόνο αν καλυφθούν οι προποθέσεις προβλέπονται από τις συνθήκες. Η πρώτη προϋπόθεση είναι στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέφερα πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο αυτή, η ενδεχόμενη προσχώρηση δεν θα πρέπει να τροποποιεί τι αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίση το πρωτόκολλο επαριθμών 8, το οποίο επιφέρει επιπλέον προποθέσει. Λέγεται στο πρωτόκολλο αυτό ότι το σχέδιο συμφωνίας θα πρέπει να διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νοσιακού δικαίου και ότι οι αρμοδιότητες επίσης των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να μείνουν ατροποποιητές και λέει επίση ότι η συμφωνία αυτή προσχώρησης δεν θα πρέπει να επηρεάζει το άρθρο 344 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παγορεύει από τα κράτη-μέλη να προβλέπουν διαφορετικού τρόπου επίλυση ζητημάτων προκύπτουν στα πλαίσια του νοσιακού δικαίου πέρα από αυτού που προβλέπονται από τι συνθήκε. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, το δικαστήριο αναφέρεται αρχικά στι ιδιαιτερότητε των συνθήκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν δημιουργήσει ένα νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα θεσμικά όργανα, στα οποία τα κράτη-μέλη έχουν παραχωρήσει μέρο τη κυριαρχία του. Ω προ αυτό το δικαστήριο λοιπόν λέει το σχέδιο συμφωνία προσχώρηση θεωρείται ασύμβατο μετά όσα προβλέπονται στι συνθήκες Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω όσον αφορά συγκεκριμένε πτυχέ. Πρώτον, υπενθυμίζει το δικαστήριο ότι ακόμα και αν η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνή σύμβαση που περιλαμβάνει δικαστικό σύστημα το οποίο μπορεί να προχωρήσει σε αποφάσεις που περιορίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι ασύμβατο με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά η αυτονομία του νοσιακού δικαίου θα πρέπει να περισωθεί. Η διατήρηση της αυτονομίας του νοσιακού δικαίου σημαίνει συγκεκριμένα ότι ένα εξωτερικό όργανο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται συνθήκες, όπως για παράδειγμα το Δικαστήριο του Στρασβούργου, δεν θα μπορεί να επιβάλλει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένη ερμηνεία του ίδιου του ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνα λοιπόν με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ελλείψεις και παραλήψεις ως προς το σημείο αυτό. Σημαντικό το κενά, διότι στη συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι θα γίνει με την διασύνδεση ανάμεσα στις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου βάσει της, του, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ε, σε εξατομικευμένο επίπεδο να προβλέπουν υψηλότερο βαθμό προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του εθνικού δικαίου, δηλαδή σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει στα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από αυτό το οποίο προβλέπεται στην ίδια τη Σύμβαση. Αυτό προβλέπεται λοιπόν για όλα τα συμβαλόμενα μέρη και συγκεκριμένα από το άρθρο 53 της Σύμβασης προκύπτει αυτό. Το δικαστήριο τώρα όσον αφορά τα κράτη-μέλη προβλέπει ότι η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βαίνει κατά της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Δεύτερον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι η αρχή της αμοιβέ εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, που είναι πολύ σημαντική όσον αφορά το νησιακό δίκαιο, δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην Συμφωνία Προσχώρησης. Στο σημείο 2 της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αποτελούν απλώς συμβαλόμενα μέρη ακόμα και προς την μεταξύ τους σχέση. Το δικαστήριο όμως ως προς αυτό μας λέει ότι αν ισχύσει αυτό το άρθρο τότε βάλετε η βασική αρχή της αμοιβέ εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα εθνικά δικαστήρια για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, το δικαστήριο αναφέρεται στο πρωτόκολλο υπαριθμών 16, πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ήδη υπογραφεί από ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρωτόκολλο αυτό, οι ανώτατε δικαιοδοσίες, τα ανώτατα δικαστήρια δηλαδή των συμβαλωμένων μερών έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμβουλευτική γνωμοδότηση όσον αφορά την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαστήριο όμω του Λουξεμβούργου θεωρεί ότι και αυτή η δυνατότητα ενδεχομένω να οδηγήσει ορισμένα κράτη-μέλη να παρακάμψουν την υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο προβλέπεται από το νοσιακό δίκαιο. Και αυτό γίνεται ιδίως αν προκύψει κάποια αμφιβολία για την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου. Τέταρτον. Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου θεωρείται το σχέδιο προσχώρησης δεν λαμβάνει αρκετά υπόψη του το άρθρο 344, το οποίο έφερα πριν από λίγο και το οποίο αναφέρεται στο πρωτόκολλο υπαριθμών 8. Διότι τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεσμεύονται να μην υποβάλλουν μία υπόθεση ερμηνεία νοσιακού δικαίου σε δικαστήριο το οποίο δεν προβλέπεται από την ένωμη τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε όμως να συμβεί στην περίπτωση της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενδεχομένως το δικαστήριο του Στρασβούργου να γινόταν το μοναδικό και πλέον αρμόδιο δικαστήριο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. και ιδίω αυτό θα προέκυπτε και μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στι διαφορέ προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρο, δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να ολοκληρώνουμε. Οι διερμηνεί δεν μπορούν να μείνουν για πάρα πολύ καιρό ακόμα μαζί μα. Θα συντομεύω, Πρόεδρε. Πέμπτον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολήθηκε και με το πρόβλημα του συνυπηρασπιστή, διότι στο συγκεκριμένο αυτό σχέδιο προβλεπόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον υπεράσπιση όσον αφορά διαδικασίες που εκδικάζονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως όταν έχουμε προσφυγή κατά κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέχει το νοσιακό δίκαιο. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αποφανθεί αν δέχεται ή όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνυπηρασπιστή, συνάγουσα στην όλη διαδικασία. Επίσης, το δικαστήριο εξέτασε τον μηχανισμό εκείνο σύμφωνα με τον οποίο το δικαστήριο θα μπορούσε να αποφανθεί εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία θα είχε αναλάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως προς αυτό, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου βλέπει ότι η Συμφωνία Προσχώρησης περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της εγκυρότητας του παραγόγου δικαίου χωρίς να δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου εκ των προτέρων όσον αφορά την ερμηνεία του παράγωγου δικαίου. Και θεώρησε λοιπόν το δικαστήριο του Λουξεμβούργου ότι αυτό παραβιάζει την αποκλειστική αρμοδιότητα που έχει για την ερμηνεία του παράγωγου δικαίου. Και τέλος, το δικαστήριο σημειώνει την ύπαρξη μιας κάποιας ασημετρίας όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου για την κοινή εξωτερική πολιτική. Ποιες είναι λοιπόν τώρα οι συνέπειες αυτής της γνωμοδότησης και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγω και στα συμπεράσματά μου κύριε Πρόεδρε. Το γνωμοδότης έχει, η γνωμοδότηση αυτή έχει άμεσες νομικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 211 σημείο 11 της συνθήκης, η συμφωνία προσχώρησης δεν μπορεί να ισχύσει με τη μορφή που έχει, εκτός και αν γίνει περαιτέρω τροποποίηση των συνθήκων ή αν τροποποιηθεί το ίδιο το κείμενο της, του σχεδίου προσχώρησης. Επομένως, η διαδικασία επικύρωσης και υπογραφής δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχιστεί. Όσον αφορά τώρα την ουσία όμως της υπόθεσης, στη γνωμοδότηση αυτή έχουμε κάποια ουσιαστικά επιχειρήματα και όχι απλά, όχι απλές λεπτομέρειες διατύπωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει μια ολόκληρη φάση περισυλλογής που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα καθήλυνα αρμόδια δηλαδή όργανα για τις διαπραγματεύσεις αυτές, να κάνουν μια αποτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχομένως και τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα καταφέρουν να αποτιμήσουν αν υπάρχει λόγος να συνταχθεί μια νέα εντολή για νέες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. θα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να δούνε αν θα μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία μια περαιτέρω απόπειρα. Τώρα, Λαμβάνοντα υπόψη τα νομικά όργανα που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, θα μπορούσε όντω να γίνει αυτή η περαιτέρω ανάλυση χωρί να τροποποιηθούν τα δικαιώματα και υποχρεώσει των κρατών μελών που αποτελούν συμβαλόμενα μέρη τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σε κάθε περίπτωση, αν λάβουν χώρα διαπραγματεύσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει ευθύ αμέσω να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα για όλα τα στάδια των εν λόγω διαπραγματεύσεων. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρέξλε, θα μπορούσατε να μας στείλετε και γραπτός τις παρατηρήσεις σας. Να τις διαβάσουν οι βουλευτές, να τις σκεφτούν και να συνεχίσουμε την συζήτηση με κάποια άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απόψε ούτε καν το 27, δεν θα συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για το σημείο αυτό είναι 2 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του κανονισμού οι τροπολογίες επίσης κατατίθενται στην Επιτροπή. Προωθούν με την ε, συνεντική διαδικασία και γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον ανατρέπουν την πρόταση του εισηγητού. Λαβερέτε αυτό παρακαλώ υπόψη σας. Και μια δεύτερη ανακοίνωση όσον αφορά το σημείο 30 γνωμοδότηση για την ε, αυτό του κ. Ντυρά. Πάλι η προθεσμία είναι 12 το μεσημέρι 2 Μαρτίου. Και η προθεσμία για τις τροπολογίες αν υπάρχουν είναι 9 Μαρτίου στο Στρασβούργο, Δευτέρα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, για τον επιπλέον χρόνο. Πέρασε συνδυάσεως.